Colleagues, uh, we'll make a start because we, we have, a, a, we have a, a busy afternoon. There are some cameras going around, but they the, the ones that are have been given permission to film for this. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει ο Πρόεδρος, ότι υπάρχουν κάποιες κάμερες, έχουν δοθεί σχετικές άδειες για την κινηματογράφηση σε συγκεκριμένες στιγμές της ε, συνεδρίασής μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης, ενημέρωση από την Europol για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της ε, Τρομοκρατίας. Ο ε, κύριο Ναβαρέτ θα καθίσει και θα μας κάνει τη σχετική παρουσίαση. Γνωρίζετε ότι από από το 2007 σε αιτήσιο επίπεδο η Europol προετοιμάζει μια έκθεση, τη ΣΑΤ ονομάζεται, η οποία δίνει την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τις τρομοκρατικές απειλές σε ολόκληρη την Ευρώπη και προετοιμάζεται τώρα η έκθεση του 2018. Ο κ. Ναβαρέτη είναι ε, υπεύθυνο είναι επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμηση τη Τρομοκρατία στη Europol και θα μα παρουσιάσει αυτή την έκθεση. <clears throat> <laughs> Έχετε το λόγο, κύριε Ναβάρετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά έχετε προσκαλέσει την Europol να σας παρουσιάσουμε μια άλλη έκθεσή μας, ακόμα μια έκθεσή μας, την έκθεση t T-SAT στην Επιτροπή Θεμελιωδών ε, Ελευθεριών. Οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της έκθεσης και πάρα πολύ σύντομα θα δημοσιοποιηθεί. Η διαδικασία είναι ε, επίπονη, είναι περίπλοκη, γιατί έχουμε ε, συμμετοχή και με συνεισφορά στοιχείων από τα κράτη-μέλη, από τη Europol, από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, προσπαθούμε να περιγράψουμε ποιες απειλές τρομοκρατικές ε, προβλέπουμε με βάση τα ε, γεγονότα του 2017. Κατά μία έννοια τι μπορεί κανείς να περιμένει τι συμβαίνει ήδη κατά τη διάρκεια του 2018 και πώς μπορούμε ή να το προλάβουμε, να το αποτρέψουμε. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά την πολέμηση τη τρομοκρατία. Πριν να μπω στην παρουσίαση τη ίδια τη έκθεση, θα ήθελα, όπω και πέρυσι, να αποτίσω φόρο τιμή σε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Φέτος 68 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις Επίσης θα ήθελα να αποτύσσω να φόρο τιμή στις διοκτικές αρχές, στις δικαστικές αρχές, στο Κοινοβούλιο, στα Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν όλοι να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Είναι μια διεθνής προσπάθεια αυτή και η συμμετοχή των βουλευτών, των κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντική για να προστατεύσουμε την ασφάλειά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω κάποια στατιστικά, αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με τις τάσεις που παρατηρούμε όσον αφορά τις απειλές της τρομοκρατίας και όσον αφορά τις προσπάθειες των κρατών μελών να την καταπολεμήσουν. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι πίσω από κάθε από, από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, την οποία πρέπει να την υποστηρίξουμε, γιατί έχασαν έναν συγγενή τους, έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο. Βεβαίω και οι δικαστέ και οι ιδιωτικέ αρχέ και οι πολιτικοί όπω εσεί κάθε μέρα προσπαθούν να κάνουν την Ευρώπη ασφαλέστερη. Ξεκινώ λοιπόν με την πρώτη μου διαφάνεια. Βλέπετε εδώ τον αριθμό των επιθέσεων. Έχει αυξηθεί το 2017. Θα προσπαθήσω να δώσω μια γενική εικόνα της κατάστασης κατά τη διάρκεια του 2017. Γνωρίζετε ότι η έκθεση T-SAT είναι αναδρομική, δηλαδή περιγράφουμε την κατάσταση την προηγούμενη χρονιά. Στο μέσο του 2018 περιγράφουμε το 2017. Έχουμε την θρησκευτική τρομοκρατία, την τζιχάντ, ίσως να μην είναι και ο καταλληλότερος όρος, Έχουμε την τρομοκρατία από αρχικές αριστερές οργανώσεις, την τρομοκρατία από αυτονομιστικές οργανώσεις και την τρομοκρατία από ακροδεξιές οργανώσεις. Ε, με αυτή την κατανομή έχουμε συμφωνήσει με τα κρατη μέλη να παρουσιάζουμε την έκθεση. Βλέπετε ότι είχαμε αναφορές σε επιθέσεις τρομοκρατικές σε 9 κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτό είναι αύξηση 45% εάν το συγκρίνει κανείς με το 2016. Όμως πρέπει να δει κανείς και τον αριθμό των θυμάτων. 68 δολοφονίες, ενώ οι δολοφονίες το 2016 ήταν 16. διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιθέσεων, ότι οι επιθέσει αυτέ είναι λιγότερο καλά σχεδιασμένε, αλλά τουλάχιστον ο αριθμός των θυμάτων ήταν μικρότερος. 107 στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά ακολουθεί η Γαλλία και μετά άλλα κράτη-μέλη. Αν εστιάσουμε τώρα στη θρησκευτική τρομοκρατία, 33 επιθέσεις είχαμε. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις γνωρίζετε ότι είναι δύσκολο ένα κράτος μέλος να αξιολογήσει ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών, έτσι ώστε να το κατατάξουμε σε μια κατηγορία. Ε, συνεχίζουμε να υπάρχουν ε, διάφορες ε, επιθέσεις, διάφορες, υποθέσεις στα κράτη-μέλη, στις οποίες να μην είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε τρομοκρατικό κίνητρο. 10 ήταν αυτές που ολοκληρώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα 62 θύματα. Όπω έλεγα, ο αριθμό των θρησκευτικών επιθέσεων είναι τέσσερις φορές μικρότερος από εκείνον των επιθέσεων με κίνητρο αυτονομιστικό. Όμως, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων είναι από αυτές τις θρησκευτικέ επιθέσεις. 62 από τους 68. Η εικόνα λοιπόν έχει αλλάξει από το 2016 και από το 2015. Βεβαίω οι διοικητικέ αρχέ, οι αρχέ συλλογή πληροφοριών, και άλλες υπηρεσίες όπως ο Όλαφ, η Europol προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλες τις πιθανές επιθέσεις, να περιμετριάσουν τις επιπτώσεις τους. Είχαμε βέβαια και μια διεθνή πραγματικότητα. Είχαμε επιθέσεις στις Φιλιππίνες, στο Αφγανιστάν, τον Ιούλιο, στην Αίγυπτο, τον Ιούλιο του στην Αίγυπτο και τον Αύγουστο στην Μπουρκίνα Φάσο. τις επιθέσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση οκτώ άτομα Ευρωπαίοι πολίτε πολίτε χωρών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχασαν τη ζωή του. Στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε ποια είναι η ε, κατανομή του αριθμού των ε, επιθέσεων σε σχέση με το κίνητρό τους. Ε, όπως σας έλεγα, ο μεγαλύτερος αριθμός των επιθέσεων ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Αύξηση λοιπόν του αριθμού των επιθέσεων όμως ήταν λιγότερο καλά σχεδιασμένες, καλά εντό εισαγωγικών και ως αποτέλεσμα ο αριθμό των θυμάτων ήταν μικρότερο συνολικά. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε την ανταπόκριση των κρατών μελών τα οποία πάντα προσπαθούν να σταματήσουν το τρομοκρατικό φαινόμενο είχαμε χίλια συλλήψεις σχεδόν ε, το 2017 975 συλλήψεις αναφέρθηκαν στη Europol ως σχετιζόμενες με την τρομοκρατία ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν ε, σχεδόν οι μισέ 365 στη Γαλλία για θρησκευτική τρομοκρατία και στις περισσότερες περιπτώσεις ε, η δίωξη ασκείται για την υποψία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά για την υποψία σχεδιασμού τρομοκρατικής επίθεσης. Επόμενο παρακαλώ. Αυτές είναι οι βασικές τάσεις που είδαμε το 17. Παρόμοιες με το 16. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση της συχνότητας, όπως ανέφερα, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν τόσο επιτυχημένη και είχαμε λιγότερα θύματα. Παρ' όλα αυτά οι τζιχαντιστές θα εστιάσω τώρα στην τζιχαντιστική απειλή, εστιάζεται σε τρεις ε, κυρίως τομείς. Ε, αδιάκριτες δολοφονίες, όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, κατά οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερε ικανότητες ή προετοιμασία. Το είδαμε αυτό ε, στο Λονδίνο τον Μάρτιο και στο Μάντσεστερ και στη Βαρκελόνη τον Αύγουστο του 2017. Επίσης, ε, σε σύμβολα του δυτικού τρόπου ζωής. Το Manchester 17 ήταν μια συναυλία pop και ε, κυρίως ε, στη Γαλλία και σε σύμβολα εξουσίας αστυνομικούς και στρατιωτικούς που φυλάνε κάποια ευαίσθητα σημεία στη Γαλλία και αλλού. Επόμενη διαφάνεια. Η βασική απειλή σχετίζεται με το λεγόμενο των ξένων μαχητών. Στρατολογούνται, ρίζοσπαστοκοποιούνται, πήγαν α, και πολέμησαν στη Συρία και αλλού. Ο αριθμός όμως αυτών των ανθρώπων μειώθηκε το 17 καθώς είχαμε μια σταθερή μείωση από το 2015 αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα πόσοι είναι αυτοί οι ξένοι μαχητές πόσους ε, κατέφεραν να σαγηνεύσουν οι τρομοκράτες, πόσοι έχουν εμπλακεί σε τρομοκρατική δράση σε Συρία και το Ιράκ και πόσοι είναι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν επιστρέψει ε, ή και στις χώρες τους. Αυτό ακριβώς τώρα προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε αυτά τα άτομα. Δεν υπάρχει ε, επίσης τρομοκρατία χωρίς προπαγάνδα. Αυτό είναι γνωστό και το γνωρίζουν πολύ καλά και οι τζιχαντιστικέ ομάδες. Η προπαγάνδα στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα είναι πολύ σημαντικά για τους τρομοκράτες για να μπορέσουν ε, να στρατολογήσουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν. Και ειδικά το Ισλαμικό κράτος έχει επιδείξει υψηλό βαθμό τεχνολογικής προσαρμοστικότητας ε, καθώς προσπαθεί να επιζήσει και να επιτύχει. Όμως, η προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους ε, υπονομεύεται από τις μεγάλες απώλειες ε, όσον αφορά την υποδομή και το προσωπικό. Προσπαθεί λοιπόν να εντείνει την διάδοση του υλικού με νέα μέσα για να έχει μια ανθεκτικότητα. Επίσης, ε, καθώς έχανε εδάφη, έχανε και μέλη ε, το λεγόμενο χαλιφάτο αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα για να ενταχθεί κάποιος στην ομάδα. Πρέπει να δούμε όμως ποιος είναι ο αντίκτυπος της απειλής από το Ισλαμικό κράτος. Ε, το Ισλαμικό κράτος αναφέρεται πλέον ε, και στον ρόλο των γυναικών. Ζητάνε από τις γυναίκες να παίξουν ένα πιο ενεργό ρόλο στη μάχη. Αυτό προωθεί και η κάιντα. Και ακριβώς ζητάνε από τις γυναίκες να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο και οι ανήλικοι, γιατί οι ενήλικοι και επίσης είναι στόχοι για την προπαγάνδα του Ισλαμικού κράτους ε, και της Αλκάιντα. Υπάρχει ε, διάδοση συγκεκριμένων εικόνων ε, ισλαμικής, ισλαμιστικής βίας στην οποία εκτίθενται τα παιδιά και βεβαίως το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό όταν δεν θα είναι πλέον τα παιδιά αυτά στα χέρια του, χαλιφά, του χαλιφάτου είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και παρά την διαδόση προπαγάνδα, φαίνεται ότι δεν έχουν καταφέρει να οργανώσουν κάποια επίθεση μέσω του διαδικτύου. Δεν λέμε ότι δεν θέλουν, αλλά χρησιμοποιούν ακόμα το διαδίκτυο για τα κοινωνικά μέσα, χρηματοδότηση, επικοινωνία. Δεν έχουμε δει ε, κάτι τέτοιο, λοιπόν, αλλά ε, παγρυπνούμε. γιατί μπορεί να υπάρχει σε απόπειρα επιθέσεων σε κράτη-μέλη. Επίσης, καθώς δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την χρήση ρόβιταχή όπλων, ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών, συντομεύεται λέει ο πρόεδρος, γιατί έχετε πολλά βλέπω. 7 λεπτά ακόμα. Έχουμε και ερωτήσεις. Η Άννα, άλλος. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, Γιατί έχετε ακόμα 8 σελίδες. Κάποιο Ο Χουάν Okay, my thesis isn't getting help by this. Um... Δεν με βοηθάτε. Πόση ώρα έχουμε. «25 λεπτά». Συνεχίστε. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Ναι, έλεγα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ρόβητα όπλων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, γίνονται έρευνες από τα κράτη-μέλη. Τα εκρηκτικά παραμένουν ε, ο προτιμόμενος τρόπος και η χρήση πυροβόλων όπλων. Έχουμε μία χρήση ε, τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, αλλά πολλές περιπτώσεις πυροβόλων όπλων σε εθνικιστική αυτονομιστική τρομοκρατία. Ε, επειδή θα απαντήσετε και ερωτήσει, λέει ο πρόεδρος. Ε, επόμενο, μάλιστα, ποιοι είναι λοιπόν οι πιθανοί επιτιθέμενοι. Το προφίλ μιλάμε για εγχώρια τρομοκρατία που ριζοσπαστικοποιήθηκε στην χώρα κατοικία χωρίς να έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό ε, πρόκειται για άτομα τα οποία είτε είναι μεμονωμένα είτε μια δεμένη ομάδα αποκτούν τις πληροφορίες και τα μέσα και προσπαθούν να επιτεθούν και μερικές φορές το κάνουν επιτυχώς. Όπως είπαμε υπάρχουν λίγα άτομα που, επιστρέφουν στην Ευρώπη από τους ε, χώρους αυτούς αλλά η αριθμή είναι χαμηλή το 2017. Μία από τις πιο σημαντικές απειλές είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί λόγω της σχέσης τους με το φαινόμενο των ξένων μαχητών. Είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, αλλά προσεχώς, ειδικά από το 2019, θα αρχίσουν να αποφυλακίζονται. Και αυτή είναι μεγάλη πρόκληση για τις υπηρεσίες πληροφοριών, για την αστυνομία, η απειλή αυτή, για να αξιολογήσουν το επίπεδο ριζοσπαστικοποίησης ή επανένταξης ε, και σοφρονισμού. Επόμενο. Σύντομα, για τους άλλους τομείς, ε, εθνικιστικές ε, και αποσχιστικές επιθέσεις συνεχίζουν να είναι περισσότερες από τις άλλες, 137 το 2017, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Ο αριθμός ε, αριστεριστικών επιθέσεων αυξήθηκε 24 ε, σε σχέση με 27 ε, για την δεξιά βλέπουμε την άκρα, την άκρα δεξιά βλέπουμε πως πέντε τέτοιες επιθέσεις έγιναν, μία είχε και ένα θύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εικόνα είναι κατακαιρματισμένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Και βέβαια υπάρχει και μια διεθνή ε, διασύνδεση και εκεί πέρα είναι ο ρόλο τη Europol. Τελευταίο. Τα κράτη-μέλη και η Europol ακριβώς προσπαθούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την έκθεση. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από όταν ε, το κέντρο μας ε, στήθηκε το 2016. Οι πόροι των κρατών μελών, στον τομέα των πληροφοριών, της αστυνομίας και κυρίως από το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν που έδωσαν στην Europol ε, τους απαραίτητους πόρους, νομίζω ότι αποδίδουν κατά την ταπεινή μου γνώμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα πρέπει ειδικά σε αυτόν τον τομέα να για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών στον τομέα της αντιτρομοκρατίας. Μάλιστα το Σάββατο είχα μια ομάδα με Ολλανδούς συναδέλφους που κοιτούσαν ε, τρία άτομα που δραστηριοποιούνταν σε Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία και εξακολουθούν να ασχολούνται με αυτό. Επίσης η προπαγάνδα ήταν ένας από τους στόχους ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τρομοκρατίας χρησιμοποιούν πάνω από 150 πλατφόρμες οι τρομοκράτες και σε συνεργασία εμείς με τον κλάδο και με τη στήριξη της Κομισιόν καταφέραμε να αναστήσουμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, του Ιντερνετ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την προπαγάνδα και η προσπάθεια στο μέτωπο της προπαγάνδας είναι σαφής. Όχι μόνο για τη διάδοση προπαγάνδας αλλά και για τα άτομα που κάνουν την διάδοση. Εδώ πέρα παίζει κέριο ρόλο η Europol. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε τα διάφορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να στηρίξουν τις ερευνές τους. Ναι, για να τελειώσω. Και τώρα έχουμε πάνω από 500.000 οντότητες ε, καταχωρήσει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών. Η τρομοκρατία είναι η δεύτερη πιο συχνή χρήση για το σύστημα αυτό και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να μειωθεί η απειλή. Γιατί η απειλή εξακολουθεί να υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν μια μείωση της απειλής από τον Οκτώβριο 17 μέχρι τον Μάρτιο 18, αλλά και πάλι είχαμε τρομοκρατικά χτυπήματα σε δύο χώρες, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Οπότε παγρυπνούμε για τα διάφορα σενάρια, εξακολουθούμε να ακούμε τα κράτη-μέλη και τι ανάγκε του. χρειαζόμαστε ακόμα τους πόρους ε, και πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτό δική σας των πολιτικών και να επαγρυπνούμε για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Τελευταία μου παρατήρηση να πω ότι οι προσπάθειες είναι πάρα πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει μεγάλες απαιτήσεις για τους υπαλλήλους ε, της Europol. Ε, ακόμα και αν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις αποφάσισαν να διαλυθούν. Το Μάιο μάθαμε ότι η ΕΤΑ που έκανε επιθέσεις ε, μετά από 50 χρόνια αποφάσισε να σταματήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΕΤΑ από το 1958 έκανε 3.300 επιθέσεις. 854 άνθρωποι δολοφονήθηκαν από την ΕΤΑ, 79 ήταν θύματα απαγωγής και 369 τραυματίστηκαν και εξακολουθούμε στην Ισπανία, στη Γαλλία πάνω από 300 ανοιχτές υποθέσεις που είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα πράγματα τα οποία διαπιστώσαμε συνάδελφοι είναι ότι δεν έχουμε μαζί μας την έκθεση TSAT. Ε, τώρα δημοσιεύεται στην TSAT συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες, ε, δίνεται η παρουσίαση και σήμερα θα γίνει δημοσίευση εκ παραλίλου. Γίνεται δηλαδή τώρα στην ιστοσελίδα της Europol ή θα βρίσκεται μέχρι το τέλος της ημέρας, αλλά δεν την έχουμε εμείς. Το λέω αυτό διότι μία από τις ερωτήσεις που μου δημιουργήθηκαν, διότι η CTC και η έκθεση TSAT και ξέρω ότι αυτοί που το παρακολουθούν το θέμα ε, σας γνωρίζουν. Ε, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για το μέλλον, μπορεί να διαφωνούν βέβαια και οι συνάδελφοι μαζί μου, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και πάλι τέτοια συνεδρίαση χωρίς την έκθεση ΤΙΣΑ. Να σας πω γιατί. Γιατί εσείς μας κάνετε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή μεν, αλλά πρόκειται για μια έκθεση η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες υπό την έννοια ότι πολλές από τις πληροφορίες που μας δίνεται για έρευνες, ε, αποκάλυψη κάποιων σχεδίων κλπ. είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Για παράδειγμα, η GCHQ στο Ηνωμένο Βασίλειο μας είπαν ότι βρήκανε τον τάδε αριθμό ε, σχεδίων. Ε, Εξορισμού βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα γιατί αυτές είναι εμπιστευτικέ πληροφορίες. Ε, για να παρακολουθούμε λίγο καλύτερα, ιδιαίτερα για τους αδέλφου οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο και παρακολουθούν λίγο πιο επισταμένα και καταλαβαίνουν τι έχει συσταθεί στη Europol και τα χρησιμοποιούν, ε, πρέπει να καταλάβουν και πρέπει να μπορέσουν να επικεντρωθούν λίγο περισσότερο στο τι ακριβώ σημαίνουν όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι σε γενικά ε, και γραμμές καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και από την Europol και από την ECTC και εκτιμούμε το έργο της Europol, αλλά θα ήθελα απλώς να σας επιστήσω την προσοχή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε πρέπει να μπορούμε να κατανοήσουμε και πώς ε, διατίθεται τα στατιστικά στοιχεία, διότι εσείς τα κάνετε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω να είναι λογικό αυτό που σας λέω. Σα το αναφέρω. Δεν είναι επίκριση. Απλώς θεώρησα ότι πρέπει να το αναφέρω. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε δηλαδή την παρουσίαση του εγγράφου με την πρόσβαση, γιατί ούτω ή άλλω είναι δικό σα το έγγραφο. Ναι, ακριβώ, γιατί αλλιώ είναι πολύ γενικά αυτά που συζητούμε. Ε, τώρα έχουμε τη δυνατότητα συνεργασία με την Europol και θέλουμε να μείνει η δομή συνεργασία. Απλώ λοιπόν το αναφέρω. Ο Χαν Φερνάντο καταρχά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πάντα σας ευχαριστώ για αυτές τις παρουσιάσεις που κάνατε και ε, για τα όσα κάνουμε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και ήθελα να κάνω μία ερώτηση την οποία θίξατε στο τελευταίο σκέλος της παρουσίασής σας. Η μη τζιχαντιστική τρομοκρατία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, ναι, υπάρχει ακόμα και αυτή τη μορφή η τρομοκρατία. Υπήρχε η ΕΤΑ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αιτίες, ε, ε, ε, εκατοντάδες δολοφονίες, αλλά η ΕΤΑ δεν είναι μόνο ένα από τα επιζώντα ήδη αυτού του πλανήτη της τρομοκρατίας. Και θα ήθελα να τονίσω τι ακριβώς γνωρίζετε εσείς, πώς αξιολογείτε τις ρίζες και τις καταβολές αυτές της μη ε, τζιχαντιστικής ε, τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών επιθέσεων που εξακολουθούν να χύνουν μην αίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μάθαμε. Για παράδειγμα, εσείς ε, ο ίδιος αναφερθήκατε σε αριστερές ή αναρχικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι υφέρπει διότι σίγουρα δεν είναι ιδεολογία. Σίγουρα δεν πρόκειται για ιδεολογία. Όπω με τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι ριζοσπαστικοποιούνται και ε, ασπάζονται τον τζιχαντισμό, θα ήθελα να ξέρω και τι γίνεται με όλες αυτές τις λεγόμενες αριστερές ή αναρχικές τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούν να καταστρέψουν το κράτος όπως ε, γινόταν στην αρχή του αιώνα. Κάποτε υπήρχε ένας τρομοκράτης που σκότωσε τον Ουμπέρτο τον πρώτο, τον ε, πρόεδρο της Ιταλίας, τον βασιλιά συγγνώμη της Ιταλίας. Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους που σκοτώνουν ε, στον 21ο αιώνα. Πρώτη μου ερώτηση αυτή. Και δεύτερον, τι διδάγματα εμείς μπορούμε να αντιλήσουμε από την αντιμετώπιση των θυμάτων. Διότι τα θύματα πάντα λένε κάτι για το τι συνέβη. Τα θύματα δεν οργανώνονται απλώς σε δίκτυα μεταξύ τους. Ορισμένες φορές τα δίκτυα αυτά ε, έχουν και σημασία όταν ε, υπάρχει ε, και οργάνωση ενός δικτύου ε, ε, ή οργανώσεις θυμάτων που υπενθυμίζουν ουσιαστικά και στις αστυνομικές αρχές και στις αρχές επιβολής του νόμου τι πρέπει να κάνουν και αυτό θα ήθελα να το σχολιάσετε αν μπορείτε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό τι μπορούν να συνεισφέρουν και σε πληροφορίες τα θύματα. Η κυρία Κινίτση παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ναβαρέτε για την παρουσίασή σας. Εσείς παρουσιάσατε ένα πολύ ε, συλλογικό πλαίσιο και αναφέρατε και μια πτυχή η οποία είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Το γεγονός ότι μειώθηκε ο αριθμός των θυμάτων σε σχέση με τις επιθέσεις και η τυπολογία των επιθέσεων που δεν είναι πλέον τόσο εξελιγμένη ε, ναι μεν έχουν οδηγήσει σε ε, λιγότερα θύματα αλλά ήταν πιο συχνές οι επιθέσεις. Όσον αφορά λοιπόν αυτή τη μορφή των επιθέσεων, ε, σε ποιο βαθμό βάσει και της ανάλυσης που έχετε κάνει εσείς ε, μπορούμε να δράσουμε προληπτικά. Δηλαδή υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι, η συνεργασία που θεωρώ ότι είναι ένας από τις θεμελιώδεις πτυχές, η συνεργασία και η ανταλλαγή των πληροφοριών. Αρκούν αυτά, είναι κατάλληλα, λειτουργούν. Κάτι ακόμα, εγώ κάνω πολύ γρήγορα πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίξατε και που σίγουρα μας ανησυχεί είναι το θέμα της επιστροφής ε, των ξένων μαχητών από τις ε, περιοχές σύραξης. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον διαπιστώνεται ότι οι τρομοκράτες έχουν βρει πιθανές διαδρομές τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να κάνουν αυτή την κίνηση και να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια ώστε να αποφύγουν και τους ελέγχους. Αναφέρομαι σε μια έρευνα που έγινε στην Ιταλία, στη χώρα μου, η οποία αξιολόγησε το ενδεχόμενο χρήσης εξωτερικών διαδρομών ε, διαδρομών οι οποίες περνάνε μέσα από τη Μεσόγειο για να μπορέσουν να επιστρέψουν στι ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μου εξοπλίστηκε για να μπορέσει να αυξήσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τη δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας ε, των πιθανών ε, επικίνδυνων στοιχείων, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν κάνετε κι εσείς κάτι σχετικό. Επίσης, το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης κάποιων, οι οποίοι βγαίνουν από τις φυλακές τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Διότι σίγουρα πρέπει να τους παρακολουθήσουμε. Το να απελευθερώνεται κάποιος από τη φυλακή δεν εγγυάται και το σεβασμό στη δυνατότητα να επιστρέψει κάποιος, ε, να ξαναριζοσκαπαστικοποιηθεί και τελικά να είναι και πιθανό ε, επικίνδυνο στοιχείο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν απατώμε πρόσφατα, είδαμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τη ριζοσπαστικοποίηση στα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον στο Βέλγιο φάνηκε ότι ήταν πολύ ψηλό ο αριθμό και θα ήθελα κάποιο σχόλιο σχετικά. Θα ήθελε κάποιο άλλο συνάδελφο, η κυρία Γκόμε, το λόγο, ναι. Κυρία Γκόμε. Καλώ ήρθατε, κύριε Ναβαρέτε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, θα έλεγα στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η Europol και η Eurojust και πώς συνεργάζεται με τις εθνικές δομές. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό και στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Εσείς πώς αξιολογείτε την επένδυση που έχει γίνει σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ρώσης παστικοποίησης, ιδιαίτερα στις φυλακές, που ξέρουμε ότι πλέον έχουν γίνει περισσότερο κέντρα ρίζοσφαστικοποίησης παρά επανένταξης και σοφρονισμού. Και επίσης σε σχέση με το ζήτημα του προσιλητισμού από ημάμιδες σε ε, φυλακές αλλά και αλλού. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι προχωράει και η χρηματοδότηση του προσιλητισμού. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξή. Προγράμματα όπω το TFTP ε, που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τις πηγές χρηματοδότησης του προσελητισμού λειτουργήσε. Τώρα, όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, όσον αφορά την ε, εξωτερική ασφάλεια, το οποίο μας το ε, επισημάνουν τη σημασία της όλοι Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν λάβει μέτρα τα οποία να βοηθούν Ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουμε ότι πολλοί από αυτούς τους ξένους μαχητές, όχι μόνο από την Ευρώπη, πηγαίνουν σε χώρες της περιοχής όπως η Λιβύη. Τρίτο ερώτημα. Τι συμβαίνει με αυτούς τους λεγόμενους μαχητές του εξωτερικού, στο εξωτερικό, που πέφτουν στα χέρια των αρχών στο Ιράκ ή σε άλλες χώρες τις οποίες θέλουν να τους ξεφορτωθούν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγυηθούν την έντιμη δίκη αυτών των προσώπων και ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη νύπτουν τα σχήρα τους και δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα για αυτούς. Μήπως αυτό είναι πολύ α, επικίνδυνο και μήπως αυτό στην πραγματικότητα ε, δεν δίνει τη δυνατότητα απόδοση τη δικαιοσύνη. Σταματάει την απόδοση τη δικαιοσύνη. Άλλο συνάδελφο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, καθυστέρησα λίγο. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλα όσα είπατε και ίσως ε, να το αναφέρατε. Σε περίπτωση όμως που δεν το αναφέρατε, θα ήθελα να ξέρω το εξής. Εσείς προσπαθείτε να καταπολεμήσετε την τρομοκρατία βεβαίως, αλλά τι, τι γίνεται με την πρόληψη. Διότι είναι καλύτερα φυσικά να προλαμβάνουμε παρά να πρέπει να θεραπεύσουμε. Είναι αυτό ε, στους τομείς δράσης σας και τι κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τερή Κάμπρας. Η κυρία Γουίμπεργκ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άκουσα απαντήσει σε πολλέ από τι ερωτήσει μου, αλλά μου περίσσεψε μία. Τι κάνετε για να καταπολεμήσετε αυτούς οι οποίοι διαμένουν παράνομα στις χώρες μας. Υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, χιλιάδες ε, άνθρωποι που βρίσκονται στις παρυφές της κοινωνίας άκουσα πολλούς κάποιον ειδικό να λέει ότι ο κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης όταν είσαι στο μπάτο της κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επίθεση στη Στοκχόλμη και η επίθεση έγινε όταν απορρίφθηκε η δεύτερη αίτηση ασύλου του δράστη. Τι κάνετε εσείς από πλευράς ε, Europol. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι σύντομα. Το είδα στις διαφάνειες, αλλά ε, η Europol νομίζω ότι είναι πολύ αντικειμενική και, και με τον προηγούμενο διευθυντή και εσείς ακολουθήσατε την ίδια άκουσα, ακολουθείτε τα στοιχεία. Αυτή η απεικόνηση Ο προηγούμενος διευθυντής πάντα πολύ προσεκτικά κοιτούσε άλλες μορφές τρομοκρατίας, γιατί μη Ισλαμική τρομοκρατία. Υπάρχει αύξηση σε κάποια από αυτές τις μορφές. Για παράδειγμα, ε, για βίαιο ακροδεξιό ε, εξτρεμισμό ε, και τρομοκρατία υπάρχει ε, καταγραφή βίαιων επεισοδίων ή είναι απλώς ε, ε, φήμες όλα αυτά. Σα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για τη δουλειά μας. Όπως σας είπα, η ΤΙΣΑ είναι απλώς μία σύνοψη της ε, δραστηριότητάς μας ε, και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής δραστηριότητας ε, και προσπαθούμε να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα για τις, κάτω, για τις χώρες μέλη για να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που διαθέτουμε για υπηρεσίες πληροφοριών, δικαστικό τομέα, αστυνομία και να μπορέσουμε να μετριάσουμε και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής έρχομαι και σε κάποιες ερωτήσεις. Εμείς ε, ασχολούμαστε με πρόληψη, με προστασία, με δίωξη και απάντηση. Ε, είναι οι τέσσερι πελάνες τη στρατηγική κατά της τρομοκρατία. Τι κάνουμε σε θέματα πρόληψη. Εδώ έχουμε δύο βασικού τομεί. Πρώτον, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι τάσει ε, των τρομοκρατών για να μπορέσουμε να δώσουμε δείξει και πληροφορίε στα κράτη-μέλη που θα μπορέσουν να τι χρησιμοποιήσουν για να προλάβουν τι επιθέσει. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε και έχουμε αύξηση των πληροφοριών τα τελευταία χρόνια, κυρίως το 2017, όπως σας είπα, ε, ενώ πριν λίγα κρατημέλη έδιναν στοιχεία, τώρα οι περισσότεροι δίνουν πολλά. Σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και μπορούμε να έχουμε περισσότερα, αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούν για πρόληψη, για ε, έγκαιρες προειδοποίησεις και να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να εξουδετερώσουμε τις επιθέσεις. Τα στοιχεία που σας έδειξα για το 2017 δείχνουν ότι είχαμε περισσότερες επιθέσεις αλλά λιγότερα θύματα. Και νομίζω αυτό διότι ε, καταλαβαίνουμε γέρος ε, ε, τα σχέδιά τους, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας με πιο ακριβή τρόπο και προλαμβάνουμε πολλά πράγματα. Επομένως, εντοπίζουμε τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να σκοτώσουν οι τρομοκράτες. Και φυσικά εργαζόμαστε και διαδικτυακά. Αναφέρθηκα στην τεράστια προσπάθεια που κάνει η Europol ή η CIRU ε, μαζί με το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους παρόχους και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζονται για να ε, μπορέσουν να διαλύσουν τον προπαγανδιστικό μηχανισμό των τζιχαντιστών. Όχι μόνο το υλικό και τις επιχειρήσεις τους, ε, αλλά και ε, τους προπαγανδιστές αυτούς αυτούς. Έχουμε ένα μηχανισμό κατά της ΑΜΑΚ ε, και βλέπουμε πώς χρησιμοποιούν τα μέσα ε, κοινωνικής δικτύωσης για να ριζοσπαστικοποιήσουν και για να τους στρατολογήσουν τελικά ως τρομοκράτες της ομάδας τους. Η προπαγάνδα σίγουρα στοχεύει σε πιο ευάλωτους ανθρώπους ε, όπως σας είπα ότι στοχεύουν σε γυναίκες, σε ανήλικους και προσπαθήσουν ε, επίσης να χρησιμοποιήσουν τα βάλιτα στοιχεία κάποιων κρατών μελών. Η ερώτησή σας κυρία μου για παράδειγμα το γεγονό ότι η παράνομη μετανάστευση ε, θέτει ανθρώπους σε πολύ ευάλωτη κατάσταση. Δεν έχουν μέσα, δεν έχουν πραγματικό τρόπο να ενταχθούν ή εύκολο τρόπο να ενταχθούν στην κοινωνία μα, επομένω είναι ευάλωτοι. Και οι τρομοκράτε το γνωρίζουν αυτό και προσπαθούν να το καταχραστούν αυτό για να μπορέσουν να λιεύσουν τρομοκράτε ε, από αυτέ τι ομάδε. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά τη, προσπαθεί να βρει τους ε, ριζοσπαστικοποιημένου και προσπαθούν να εντοπίσουμε και αυτού που ε, στρατολογούν ε, είτε στο διαδίκτυο είτε διαζώσεις για να μπορέσουν να αποφύγουν να συμβεί κάτι τέτοιο σε κάποιες χώρες. Έχουμε κάποια παραδείγματα παρανόμων μεταναστών που τελικά βρέθηκαν στην Ευρώπη, ριζοσπαστικοποιήθηκαν και ε, δυστυχώς έκαναν και κάποια πράγματα τα οποία είχαν θύματα ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομία επικεντρώνεται στην πιο βίαιη πτυχή, αλλά βέβαια και η κοινωνία θα πρέπει να κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες κατά την άποψή μου ε, για να μειώσουν τις συνέπειες της στρατολόγησης, της ριζοσπαστικοποίησης και τελικά και των τρομικροετικών επιθώσεων που σχετίζονται με αυτούς ευάλωτες τομείς της κοινωνίας μας που ε, βρίσκονται στις περιοχές μας. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους αποφασίζουν να ε, ε, γίνουν τρομοκράτες. Και ε, λέμε γιατί ήταν τόσο σημαντικό να γίνουμε μέλη της Αλκάιντα του Ισλαμικού κράτους. Έχουμε περίπου χίλιους Ευρωπαίους πολίτες, κατοίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν να ενταχθούν στους κόλπους του, του Ισλαμικού κράτους και της, και της Αλκάιντα. Ε, έχουμε ανθρώπους που πηγαίνουν και στις περιοχές σύραξης ε, και πριν το 2013 και μετά το 2013 οι τελευταίοι έλαβαν και στρατιωτική εκπαίδευση ε, και είναι και επικίνδυνοι. Ίσως οι τελευταίοι που πήγανε στη Συρία έχουν τελείως διαφορετική ε, νοοτροπία και κάτι άλλο στο μυαλό τους. Και ε, έχουμε πει ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν είναι πλέον ομοχλός κίνησης. Υπάρχει, το χρησιμοποιούν, χειραγωγούν την περιοχή, ώστε να ε, υπάρχει το δέλεαρ να ενταχθούν στο Ισλαμικό κράτος, αλλά υπάρχουν και πολλοί προσωπικοί λόγοι, εκδίκηση. Κάποιοι από αυτούς σε πολλές φορές, ε, ε πάσχουν και από ψηφικικές διαταραχές. Ε, για να μπορέσουν ορισμένες φορές να διεκδικήσουν τα προσωπικά τους θέματα εντάσσονται στο Ισλαμικό του κράτος. Τώρα για τους υπόλοιπους. Έχουμε και κάποιους τρομοκράτες οι οποίοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ε, οδούς μετανάστευσης ε, για να ε, προχωρήσουν και να προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Ιταλία και την Ελλάδα στα hot spots. Γίνονται εκεί έλεγχοι σε δεύτερο βαθμό και ε, βλέπουμε συστηματική χρήση των τρομοκρατών από, αυτούς τους ε, από αυτές τις οδούς, αλλά είμαστε πολύ δραστηριοποιημένοι και κάποιοι από εσά ε, είπατε αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποιους οι οποίοι ήταν εγκληματικά στοιχεία και ριζοσπαστικοποιούνται στη φυλακή, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν για συνωμοσία, για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ομάδες και μετά ε, μετά από την έκτηση της ποινή τους ε, θα αφαιθούν ελεύθεροι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούμε. Ε, προσπαθούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα για να καθορίσουμε ένα προφίλ, να μπορούμε να κάνουμε κατάλληλη αξιολόγηση και να προτείνουμε στα κράτη-μέλη να έχουν κάτι για πρόληψη αλλά και για αντίδραση. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα ε, να ε, μα βοηθήσουν για να του βοηθήσουμε κι εμείς για να δούμε τι πιο πιθανέ απειλέ και να μπορέσουμε να μετριάσουμε το ενδεχόμενο τρομοκρατική απειλή. Υπάρχει κάποια συνεργασία ε, σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, σε διάφορου τομεί, αναφέρθηκα στην πρόληψη. Και το τελευταίο που θα αναφέρω είναι η μη Ισλαμιστική τρομοκρατία, πολύ συχνά μη τζιχαντιστική τρομοκρατία, την οποία ανέφεραν κάποιοι από εσά. Χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία για να καθορίσουμε ένα φαινόμενο. Είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι τρόπον την αποδεκτή και πάντα μπορούμε να την ε, υπερασπιστούμε, αλλά υπάρχουν ε, ε, διάφορα θέματα. Ε, τζιχαντιστές, αποσχιστικές τάσεις, αριστερή, δεξί και έχουμε δει ιδίω σε αριστερά, αριστερή μορφή προτρομοκρασίας και κάποιες μορφές ε, ε, τρομοκρατίας. Αλλά αυτή η αντισυστημική τρομοκρατία που είχαμε στη Γερμανία σε κάποιες περιοχές του Αμβούργου ή και στη Γαλλία είναι πολύ ανησυχητική. Τα κράτη-μέλη που καταγράφουν τέτοια στοιχεία που έχουν τη η πτυχή ε, κάποιων συγκεκριμένων ομάδων και δεξιών και αριστερών προσπαθούν να μειώσουν το ενδεχόμενο περισσότερης βίας ε, και επιθέσεων. Ε, είναι χαμηλές αυτές οι πιθανότητες, αλλά θέλουμε να τις κρατηρήσουμε όσο πιο χαμηλές γίνεται. Και κάτι τελευταίο. Ο στόχος είναι πάντα χειραγώγηση. Προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινωνία, το πολιτικό περιβάλλον και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τους δελεάσουν, να ριζοσπαστικοποιηθούν και να ενταχθούν στους κόλπους τους. Έχουμε πάρα πολλέ ε, ε, μελέτες για τη ε, τζιχαντιστική ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε βρει ε, τα εργοστάσια παραγωγή, αν θέλετε, τα υπέρ και τα κατά. Και έχουμε και αποσχιστική ριζοσπαστικοποίηση, αριστερή, δεξιά ριζοσπαστικοποίηση. Ε, χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε για να δούμε τα προφίλ, αλλά δεν απέχουμε και πάρα πολύ και θέλουμε να ξέρουμε και την κοινωνική πτυχή, αλλά και την νομική πτυχή. Κατά βάση όμως θέλουμε, ε, ε, έχουμε χειραγώγηση και μια ε, τη αντισυστημική απάντηση που χρησιμοποιεί τη βία ως εργαλείο για να αλλάξουν οτιδήποτε θέλουν να αλλάξουν στις κοινωνίες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά βέβαια έχουμε και άλλα δύο πολλά σημαντικά θέματα. Γνωρίζουν σήμερα επίση οι συνάδελφοι ότι έχουμε το αυστηρό όριο του να έχουμε τελειώσει μέχρι τι 6.30 και για λόγου διερμηνία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σύντομα, εξάλλου, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή τη Europol. Καλή επιτυχία στο έργο σα και σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ. Ο... Καθώς φεύγει ο κύριος Ναβαρέτη θα ζητήσω από τον διευθυντή τη υπηρεσίε θεμελιωδών δικαιωμάτων έρθει. Συνάδελφοι, για λόγου που δεν γνωρίζω, έχουμε μόνο 45 λεπτά στη διάθεσή μα για το επόμενο θέμα. Είναι μια κοινή συζήτηση για την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Τέρι Κάμπρας, είναι παρόν. Θα παρουσιάσει την προσχέδιο έκθεση του μετά τις δύο παρουσιάσεις που θα ακούσουμε. Όπως σας είπα, μόνο 45 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Φλάχαρτη, ούτε το το F. Ελπίζω στην επόμενη επίσκεψη σα να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα να σας ακούσουμε. Σε κάθε περίπτωση μπορώ ήδη να σα συγχαρώ για το έργο της ε, υπηρεσίας σας που είναι εξαιρετικό. Ναι, λοιπόν και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας παρουσιάσετε συνοπτικά την ετήσια εκθεσή σα και μετά θα έχουμε κάποιες ε, ερωτήσεις από τα μέλη και πάλι να σας ευχαριστήσω για το έργο της υπηρεσίας σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας προσωπικά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεγάλο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει στο έργο της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων καθ' όλη τη ε, δράση μας. Ε, θα σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση 2018, η οποία βέβαια αναφέρεται στις εξελίξεις το 2017. Έχουμε 10 κεφάλαια τα οποία πάνω κάτω αντιστοιχούν στο πολιετές πλαίσιο με το οποίο μας έχει πρικήσει ο νομοθέτης. Θα δείτε ότι στην έκθεση γίνεται μια πολύ λεπτομεριακή ανάλυση και από την πλευρά του Διευθυντή και της α, Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά επίσης και μέσω του δικτύου FRANET, του δικτύου των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουμε στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να δούμε τι λειτουργεί, ποιο, που είναι, είναι τα προβλήματα, αλλά επίσης και πώς μπορούμε να έχουμε πρακτικές οι οποίες ε, να είναι βέλτιστες. Και καταλήγουμε σε κάποιες συμπεράσματα και σε κάποιες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και προς το Κοινοβούλιο, που είναι η άποψη της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πώ θα μπορούσαμε να ενισφέρουμε στο έργο σα. Ε, Μια και δεν έχω πολύ χρόνο στη θέση μου, θα σας δώσω μόνο ορισμένα στοιχεία, πολύ συνοπτικά. Ας δούμε, πρώτα το ζήτημα της εφαρμογής του θεμελιώδους χάρτη ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως και προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει μια μικρή ε, βελτίωση σε εθνικό επίπεδο, μικρή. Βλέπουμε κάποιες ε, παραπομπές να γίνονται στην, στη θεμελιώδη χάρτη στα δικαστήρια και στο κοινοβούλιο, αλλά όχι επαρκής αριθμό είναι ευθύνη και δέσμευση των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους να προωθούν τη χρήση του, της θεμελιώδους χάρτας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στι γενικέ γραμμέ πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει σύγχυση όσον αφορά την εφαρμογή ε, του χάρτη, ιδίω ε, σε σχέση με το εάν ένα ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Για αυτόν τον λόγο έχουμε προσπαθήσει μέσω γνωμοδοτήσεων να ε, καταστήσουμε πιο γνωστή, περισσότερο γνωστή τη χάρτα και ιδιαίτερα στο διασυνοριακό επίπεδο. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προσπαθεί να συνεισφέρει. Τις επόμενου μήνες θα δημοσιοποιήσουμε ένα εγχειρίδιο για το πώς μπορεί να χρησιμοποιείται ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κρατη σε εθνικό επίπεδο. Το εγχειρίδιο αυτό θα απευθύνεται στους βουλευτές. Επίσης έχουμε ξεκινήσει να στείλουμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό κατάρτιση προς τις Εθνικές Επιτροπές Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, έτσι ώστε εκείνε να αξιοποιούν ε, τον χάρτη στο έργο τους. Μετά. Όπως γνωρίζετε δεν είναι μόνο μεγάλη προτεραιότητα για εσάς αλλά και για μεγάλη προτεραιότητα για την ε, υπηρεσία ανθρωπίνων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων διάφορες διάφορα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε εκθέσεις για την κατάσταση επιτόπου για 14 κράτη-μέλη όσον αφορά το μητράστης και το άσυλο, 14, ανάμεσα στα οποία η Ιταλία και η Ελλάδα. Έχουμε προσπαθήσει μέσω προγραμμάτων κατάπτυσης να συνεισφέρουμε και επίσης μέσω νομικών γνωμοδοτήσεων. Το Δεκέμβριο δημοσιοποιήσαμε μια έκθεση που εντοπίζει πέντε ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, στον τομέα της μετανάστευσης. Πρώτα απ' όλα, δυσκολία στο να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε κάποια κράτη-μέλη, στο να υποβάλει μια αίτηση ασύλου και να εξεταστεί. Βεβαίως, πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτά τα προβλήματα εκφράζονται και λαμβάνουν υπόσταση πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Δεύτερο πρόβλημα. Σε κάποια κράτη-μέλη είτε οι πρωτοβάθμιες είτε δευτεροβάθμιες διαδικασίες ασύλου είναι ε, προβληματικές. Είτε από πλευρά διαδικασία είτε από πλευράς ε, διάρκεια. Τρίτον, προβλήματα όσον αφορά τι υποδομέ στι οποίε στεγάζονται οι ε, ετούντε άσυλο Τέταρτον, έχουμε συστηματικά προβλήματα με τους ε, ανήλικους ετούντε άσυλο, με διαφορετικό τρόπο αυτό από χώρα σε χώρα και τέλος υπερβολική χρήση της κράτηση ω μέτρου και συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης παιδιών σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες χώρες. Το συμπέρασμα από αυτά τα ευρήματα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ουσιαστικό πλαίσιο για να παρακολουθούνται οι απελάσεις από πλευρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρώτον. Και δεύτερον, κατά τη διάρκεια του 2017 η υπηρεσία μας ε, ε, εξέτασε αυτές τις υποθέσεις πολύ διεξοδικά. Και δεύτερον, πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν τα μεγάλα πληροφοριακά συστήματα και ιδιαίτερα η διαλειτουργικότητα που αρχίζει να αναπτύσσεται των πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο των συνόρων, τι επιπτώσεις θα έχει στα ανθρώπινα δικαιώματα και για αυτό το θέμα έχουμε δημοσιοποιήσει διάφορες γνωμοδοτήσεις. Συνολικά μιλώντας για το ζήτημα της μετανάστευσης, μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η υπηρεσία μας θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα πάρα πολύ συστηματικά και στο μέλλον. Μιας και μίλησα για μεγάλα πληροφοριακά συστήματα, έρχομαι και στο γενικότερο ζήτημα της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ραγδαία ε, εξέλιξη και κατά τη διάρκεια του 2017 της πληροφορικής αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Είναι μια θετική αλλαγή στις κοινωνίες μας που μας δίνει πολλές δυνατότητες για πάρα πολλά πράγματα από την παροχή υγείας ε, μέχρι τις κοινωνικές σχέσεις. Όμως οτιδήποτε έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις θετικές μπορεί να έχει και μεγάλους κινδύνους. Τους κινδύνους αυτούς προσπαθούμε να επισημάνουμε στην έκθεσή μας καλωσορίσαμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017 να προσπαθήσει να κατεβάσει ιστοσελίδες που ε, προσπαθούσαν να διαδώσουν ε, τη ρητορική του μίσους. Καλωσορίσαμε επίσης την θέση σε εφαρμογή του, κανονισμού, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, σε ορισμένα αναπτύχθηκαν ε, εθνικές πρακτικές τις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Στο μέλλον, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα συνεχίσει να ασχολείται ουσιαστικά με το θέμα και έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της τεχνικής της νοημοσύνης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ελπίζω στις αρχές του 19 να μπορούμε σύντομα να σας ε, ενημερώσουμε σχετικά για ερωτήματα όπως για παράδειγμα πώς φροντίζει κανείς ότι ένας αλγόριθμος σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή πώς μπορεί να εξασφαλίσει ότι στην τεχνολογία blockchain που γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να διαγραφεί από, την, από το σχεδιασμό της τεχνολογίας, πώς μπορεί αυτό να είναι συμβατό με το δικαίωμα στη λύθη. Δυστυχώς, το 2017 είχαμε πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο διακρίσεων ε, σε πολλά κράτη-μέλη. Θα θυμάστε ότι το 2017 δημοσιοποιήσαμε στοιχεία συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη εκτός δύο ε, που αφορούσαν στις διακρίσεις που υφίστανται μια σειρά ε, πολλές μειονότητες. Πρώτα απ' όλα για εκείνους που δηλώνουν ε, μουσουλμάνοι, την κατάσταση των Ρωμά, την κατάσταση των Εβραίων. Ιδιαίτερα μιλώντας για τους Ρωμά, αυτό που διαπιστώσαμε το 2017 ή μάλλον αυτούς το οποίο προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στο 2017 ήταν η αύξηση του αισθήματος ε, κατά τον Ρωμά, το αντιαθηκανισμού. Ε, Μιλώντας γενικότερα τώρα για το ζήτημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό και το βρίσκουμε ξανά και ξανά στις μελέτες μας, ότι χρειάζεται μια οριζόντια προσέγγιση, δηλαδή. Ε, ε αυτό το βλέπουμε ακόμα περισσότερο στο ε, ζήτημα των γυναικών Δηλαδή, ακόμα και εντό των διακρίσεων, οι γυναίκε μουσουλμάνε υφίστανται ακόμα μεγαλύτερε διακρίσει από του άνδρε μουσουλμάνου. Οι γυναίκε Ρωμά ακόμα μεγαλύτερε από του άνδρε Ρωμά. Τα αποτελέσματα, τα ευρήματα της μελέτης μας καταδεικνύουν ότι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι κοινότητε αυτές που πέφτουν θύμα διάκριση σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Δεν γνωρίζουν ότι οι ορισμένες συμπεριφορές, οι πολιτικές τις οποίες υφίστανται είναι ε, μη αποδεκτές, είναι λανθασμένε, είναι παράνομες. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε το έργο μιας ομάδας εργασίας που προσπαθεί να συλλέγει στοιχεία για τη ρητορική του μίσους και σύντομα θα έχουμε μια έκθεση από αυτούς. Επίσης θα ξεκινήσουμε μια συγκεκριμένη μελέτη για τον αντισημιτισμό και θα ε, προσπαθήσουμε πλέον να, να κοιτάξουμε και άλλες ομάδες όπως για παράδειγμα να, εξετάσουμε την κατάσταση των Αφρικανών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζουμε και ένα εγχειρίδιο σε σχέση με ε, αστυνομικές πρακτικές που είναι από τη φύση τους ε, εισάγουν διακρίσεις όπως για παράδειγμα το profiling. Κάθε διάρκεια του 2017 συνεχίσαμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας για ορισμένες καταστάσεις, ορισμένα μοτίβα και καλωσορίσαμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε έμφαση και μέσω του συνεδρίου της ε, στα δικαιώματα των γυναικών. Είναι όμως σοκαριστικό να, να βλέπει κανείς ότι στα συμπεράσματα ε, χρειάστηκαν δύο σελίδες για να μιλήσουμε για το φαινόμενο της, ε, των δολοφονιών γυναικών και κοριτσιών. Αυτό στην Ευρώπη, στις μέρες μας. Έχουμε επίσης επιλέξει ως θεματικό ε, κεφάλαιο, ως θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το 2018, την προσέγγιση ανθρω... τους γύρανσης από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό το κάνουμε γιατί διαπιστώνουμε ότι έχει, έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διακρίσεις ε, των οποίων ε, πέφτουν θύματα οι ηλικιωμένοι πολίτες. Διαπιστώνουμε ότι από το Ευρωβαρόμετρο οι διακρίσεις κατά των περισσότερων ηλικιωμένων, των ηλικιωμένων είναι η πιο διαδεδομένη μορφή διάκρισης στις κοινωνίες μας. Και πάλι οι γυναίκες ε, πλήττονται περισσότερο από τους άνδρες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το, η σύνταξη ενός άνδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 37% υψηλότερη από αυτή μιας γυναίκας. Βεβαίω εστιάζουμε σε αυτό το θέμα γιατί είναι σοβαρό θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίση και εξαιτία τη γύραση του πληθυσμού στην Ευρώπη, τη δημογραφική εξέλιξη στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι θα, θα είναι όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Και ζητάμε μέσω του κεφαλαίου Focus να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα στα εθνικά επίπεδα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να γνωρίζουμε δηλαδή την διάσταση της ηλικία σε οποιοδήποτε ζήτημα μπορείτε να φανταστείτε και όσον αφορά την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλωσορίζουμε την ανάγκη για μια μόνιμη εστίαση στι ανάγκε των ηλικιωμένων, στον πυλώνα παραδείγματο χάρη ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην εστίαση που απαιτείται όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ε, ίσης μεταχείρισης. Τελειώνω εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και να πω πως όλες οι γνωμοδοτήσεις της έκθεσης είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο σε όλες τις ε, γλώσσες και η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Μάικλ. Βλέπω εδώ πέρα είναι και ανακυκλώσιμο. Το πρόσκυσα δεν είναι από το άλλο το χαρτί. Ωραία, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βλησιάζει ε, πέντε και... Ναι, τα ξέρω, έχουμε μετά άλλο θέμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ε, Κριστίν. Ναι, η παρέμβασή μου περισσότερο ήταν ε, ε, προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις ε, εκθέσεις σας. Προς τον κύριο Κράμπιτ, λοιπόν, τρεις ερωτήσεις. Όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων, η Επιτροπή στην έκθεσή της χαίρεται και εμείς επίσης, συγγνώμη Κριστίν, μισό λεπτό, δεν δουλεύουν τα ακουστικά ο διευθυντής του FRA χρησιμοποιήσει τα ακουστικά κάποιου άλλου και ασχολείται και με ψηφιακά ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα σχολιάσω καν. Euh, euh, για την έκθεση λοιπόν ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρώτο σημείο αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου. Χαιρόμαστε όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 για την Πολωνία, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι είναι μακρά ακόμα η πορεία, αλλά επίσης ε, και για την Ουγγαρία η οποία ε, δεν εφαρμόζει σωστά την νομοθεσία σε θέματα μετανάστευσης ε, και ασύλου, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει και να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7 και για την Ουγγαρία. Γιατί δεν ξεκίνησε. Όσον αφορά το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών, βλέπουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση στην έκθεσή σας ότι οι επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών αναφέρονται ε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ ανησυχητική οπισθοδρόμηση και κυρίως αναφέρομαι στα σεξουαλικά και αναπορικογικά δικαιώματα και μάλιστα αυτό ε, θα έπρεπε είναι, να είναι στο επίκεντρο των θεμάτων του 2018 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερο όσον αφορά το χάρτη. Θα μπορούσαν να προσθεθούν αυτά τα δικαιώματα στο χάρτη. Προβλέπεται αναθεώρηση του χάρτη για να συμπεριληφθούν και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή προστασία των γυναικών σε αναποριαγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι τελευταίο το οποίο ίσως ε, θα βελτιώσει λίγο την κατάσταση. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα κάνει για την, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα και την οδηγία συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματική ζωής, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε όταν το Συμβούλιο φαίνεται να προσπαθεί να ε, υποσκάψει την ε, πρόταση ε, της πραγματικής εναρμόνισης και προσπαθεί να περάσει σε μία συμφωνία ανακράτος μέλος την οποία, η οποία τορπιλίζει τα όσα προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, κοιτάξτε, έχουμε 7 ομιλητές και η Κομισιόν θα κάνει και αυτή η παρουσίαση και μετά. Πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Κράμπιτ. Σε 20 λεπτά όλα αυτά. Εντάξει, είπαμε, είμαι μάγος, αλλά... Λοιπόν, κύριε τερικάμπρασκο. κούκου, δύο λεπτάκια, παρακαλώ, για να τελειώνουμε μέχρι τις 5 αυτό το θέμα. Δύο λεπτά για όλους. Συναντιόμαστε ξανά, αγαπητέ. Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι αυτό το οποίο λέτε ότι δεν γίνονται αρκετές ε, προσπάθειες για να προωθηθεί η χάρτα στα κράτη-μέλη της Ένωσης στο εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι συγκλονιστικό γιατί δεν είναι θέμα χάρτας της Ένωσης. Αυτές είναι οι βασικές αρχές οποιοδήποτε δημοκρατικού κράτους στην Ένωση. Αν έχουν αυτές τις αρχές στα συντάγματα, που είναι δυνατόν να υπερασπίζονται αυτά τα συντάγματα και όχι τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εάν ε, μπορείτε να Μα το διευκρινίσετε αυτό, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Πίτερ Νίντερ Μιούλα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά έχω να αναφέρω δύο πράγματα. Βλέπουμε τεράστιε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών για το θέμα των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη που σε κάποιους ε, τομείς έχουν διαφορές, αλλά έχουμε κάποια κράτη-μέλη όπου η βία στα θέματα αυτά φαίνεται ότι είναι πρακτική κυβερνητική. Ότι είναι η βάση δηλαδή της ε, πολιτικής διακρίσης, ε, ρητορική κτλ. Πώς το βλέπετε αυτή την κατάσταση δηλαδή που αλλάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να μιλήσω για συγκεκριμένους ε, τομείς, ε, για τη βία, αλλά να χρησιμοποιείται η βία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βάση για την πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πίτερ, ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Και για την έκθεση και για τα ευρύτερα ζητήματα ζητώ συγγνώμη. Τώρα τι να κάνουμε. Αυτό τον χρόνο έχουμε. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, το κύριο Φλάχερτη για τα όσα κάνει και για την έκθεση. Εγώ αυτή τη φορά έχω μία ερώτηση για την Ιταλία και την ε, μεταχείριση των Ρωμά στην Ιταλία, ε, την οποία βρίσκω ιδιαίτερα ανησυχητική. Η τελική κυβέρνηση μέσου του Υπουργού της Εσωτερικών είπε τις προηγούμενες ημέρες ότι δυστυχώς πρέπει να ε, ε, παρακολουθούμε τους Ιταλικούς ε, Ρωμά και με αυτό υπονόησε ότι οι υπόλοιποι, οι μη Ιταλοί, με ευρωπαϊκό διαβατήριο θα πρέπει να φύγουν. Και νομίζω ότι κάνετε μια έρευνα για την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη και θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό δυσκολεύει τη δική σας τη δουλειά σε θέματα συνεργασίας με ε, Ρωμά, διότι ένα τμήμα αυτό το Ρωμά ε, θα κρυφτεί οι νομάδες και δεν θα συνεργαστούν. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την ανακοίνωση ε, για την ε, καταστροφή των ε, καταβλισμών στο Ρωμά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ιταλία, αλλά κάθε φορά παρουσιάζεται ο σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν αυτοί οι καταβλισμοί. Αλλά υπάρχει τέτοια ε, σύσταση. Το ρωτάω και την, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η σύσταση γίνεται βάσει των συγκεκριμένων συνθήκων. τι γίνεται με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, καταστρέφεται ένας καταβλισμός όταν προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση σε αυτούς που μένουν σε καταβλισμούς. Ε, ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, Μπίρκη Τσίπελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πολλές σημαντικές ερωτήσεις, οπότε δεν θα μιλήσω. Ευχαριστώ, Μπίρκητ. Άννα Γκόμες, ε, σύντομες να είστε, παρακαλώ. Ναι, η ερώτησή μου αφορά ακριβώς το νέο περιβάλλον με τα κοινωνικά δίκτυα και την κοινωνία των πληροφοριών. Να λέτε για τις συνέπειες των ε, μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ποιες συνέπειες βλέπετε από την σκοπιά της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης, γιατί μπορεί να είναι ακόμη πιο ολοκληρωτικό το πράγμα, το αποτέλεσμα με τα μαζικά δεδομένα. Ναι, ναι, ένα τεράστιο θέμα στο οποίο μπήκατε. Κατερίνα Τσινίτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ, κύριε Φλάχερτη. Ε, δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκε με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα δικαιώματα των ανηλίκων ασχολείστε για παράδειγμα με το θέμα της ε, ε, φτώχειας που είναι και οικονομική ε, και ηλική αλλά και εκπαιδευτική ένδυα. Θα ήθελα να ρωτήσω στη σχέση μεταξύ ανηλίκων και διαδικτύου που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουν γνώσεις οι νέοι, για να κοινωνικοποιηθούν κλπ. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε από τους κινδύνους, από το ε, cyber bullying ε, για παράδειγμα ή τους εκβιασμούς που ε, μπορεί να δημιουργήσουν σε δραματικά προβλήματα για τους ανήλικους. Επίσης, το άλλο θέμα είναι η βία κατά των γυναικών. Είμαστε μία από τις χώρες οι οποίες προσυπέγραψαν αμέσως τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, κυρώσαμε τη σύμβαση και μετά την περάσαμε στην ποινική μας ε, νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, οι γυναικοκτονίε εξακολουθούν να είναι πολύ αυξημένε στον αριθμό. Και επίση, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε ε, και τι γυναίκε. Ε, το φαινόμενο, ναι, μεν υπήρξαν παρεμβάσει, αλλά συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανεί. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω, Μάικολ, και να τονίσω στα μέλη ότι πέραν της έκθεσης υπάρχει και δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί σας αν θέλουν κάτι συγκεκριμένο. Θα ήθελα να το τονίσω στους συναδέλφου που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τη δουλειά του. Έχετε κατά νου λοιπόν αυτό, διότι υπάρχουν μέλη που ακόμα δεν έχουν επικοινωνήσει. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και αν θέλετε απαντήστε στις ερωτήσεις. Θα απαντήσω τις ερωτήσεις που απευθυνθήκαν σε μένα τα υπόλοιπα της κυρίας Μπονεφού νομίζω απευθύνθηκαν προς την ε, Κομισιόν. Να απαντήσω στον κύριο Τερικάμπρας και την ε, παρατήρησή σας ε, του ότι δεν γίνεται κάποια κίνηση για να προωθηθεί η χάρτα. Για να μην υπάρχει αίσθηση της πλήρους καταστροφής βεβαίως δεν θέλω να υπονοήσω ότι τα κράτη-μέλη δεν προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κάνουν. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη που έχουν ε, εθνικά σχέδια δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά κανόνα όμως ε, βασίζονται στην ε, ΕΣΔΑ και σε συμβάσεις του ΟΗΕ όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οπότε απλά το συγκεκριμένο μέσο, η χάρτα, φαίνεται ότι δεν έχει προσελκύσει την προσοχή που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική να επιτευχθεί. Αυτό είναι αν θέλετε συμφωνώ με τον κύριο Νίτερ ότι έχουμε ένα φαινόμενο κάποιων πολιτικών που αμφισβητούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα έλεγα ότι εμείς φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων είμαστε ένα μικρό κομμάτι της αντίδρασης σε αυτά τα πράγματα που είναι βεβαίως τελείως πολιτικά. Και το ερώτημα είναι τι θα πρέπει να κάνει ένας φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος ε, είναι νόμος. Να επιμείνουμε σε αυτό, να μην είναι κάτι επιλογή. Δεύτερον, να μιλάμε για τις παραβιάσει. Τρίτον, με βάση δεδομένα κάτι για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Τέταρτον, πρέπει να ε, μεταφέρουμε καλύτερα τα μηνύματά μας και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ακριβώς να λέμε γιατί λέμε κάποια πράγματα δεν είναι κάτι το ενάρετο και καλό, οδηγούν σε καλύτερη κοινωνία και πρέπει να έχουμε ε, μεγαλύτερη επαφή με το ευρύ κοινό. Το ευρύ κοινό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τέλος πρέπει να οικοδομήσουμε νέες συμμαχίες για να προωθήσουμε μια κοινωνία που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μεγάλη ενέργεια στις ε, κοινωνίες μας ε, που δεν έχει ακριβώς διοχετευτεί κάπου για αυτά τα ζητήματα. Αναφέρατε κυρία Σπινέλη το θέμα των δηλώσεων υπουργών. Οπωσδήποτε ανησυχώ ε, για κάτι το οποίο ακριβώς θα μπορούσε να γίνει ε, αλλά περισσότερο για αυτά τα οποία λέγονται, κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των Ρωμά προς τα μας και θα έπρεπε η Ιταλική κυβέρνηση να γνωρίζει το ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσει περισσότερα δεδομένα για τους Ρωμά για να προστατεύσουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα και οπωσδήποτε θα παρακολουθήσω αυτό το ζήτημα, η υπηρεσία δηλαδή. Κύριε Γκόμες. Ναι, δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για την δουλειά που κάνουμε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των μαζικών δεδομένων. Το μήνυμα είναι ε, σαφές. Ε, έχουμε ε, περάσει πλέον αυτό το σημείο γιατί είναι τα δεδομένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας ε, και δεν γίνεται αλλιώς. και δεν έχω να πω κάτι πέρα από το ότι ο οδηγός του profiling ακριβώς ε, θα θέσει το ζήτημα των αλγορίθμων και της διακριτικής μεταχείρισης. Και τέλος κυρία Κινίτσι. Αντιλαμβάνω πλήρως αυτό το οποίο λέτε για την προστασία των παιδιών, ε, κύβερνο, τσαμπουκάδες και πορνογραφία. Και βεβαίως ακριβώς ε, το θέμα εδώ πέρα είναι η περική προστασία, η προστασία των παιδιών, αλλά δεν είναι κάθε πτυχή αυτού του θέματος ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά όπου μπορούμε να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε. Για τη βία κατά των γυναικών ε, θα συνεχίσουμε Βεβαίω να ενθαρρύνουμε την κύρωση τη συνθήκη Κωνσταντινούπολη ακόμα δεν έχει κυρωθεί, οπότε δεν έχουμε ακόμα την νομοθεσία, την έχει υπογράψει αλλά δεν έχει κυρώσει ακόμα την ε, Σύμβαση Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπογραφή μια συνθήκη βεβαίω δεν είναι το τέλο του προβλήματο. Κατόπιν γίνονται όλε οι προσπάθειες για να αλλάξουν οι προκαταλήψεις στην κοινωνία και εδώ πέρα είναι ο δικός μας ο ρόλος. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο ακόμα σε σχέση με το τι νομίζαμε πριν από λίγα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σύντομος. Ε, υπήρχε ερώτηση για την Ιταλία, την απαντήσατε, την απαντήσατε μάλιστα. Ε, την απάντησα όπως μπορούσα. Μπάρμπαρα. Ναι, είχα ρωτήσει επίσης αν υπάρχει κάποια ένδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να ε, προτείνει ε, τον, ε, την καταστροφή των καταβλισμών Ρωμά. Γιατί στην Ιταλία λέγεται συνεχώς ότι η Ευρώπη μας ζητά να καταστρέψουμε αυτούς τους καταβλισμούς. Δεν αποφεύγω την ερώτηση. Νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει καλύτερα από μένα. Ο Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση δεν έχει πει σε κάποιον να καταστρέψει ένα καταβλισμό. Ευχαριστώ. Και βέβαια δεν ε, τη βοηθάει το γεγονό ότι δεν είχαμε καθόλου χρόνο για το θέμα αυτό. Έπρεπε να τα είχα προβλέψει κάποια θέματα, ειδικά όταν ο Πίτερ ε, ε, έχει τόσε πολλέ ερωτήσει να απαντήσει. Δεν βοήθησε. Και πραγματικά λυπάμαι που δώσαμε μόνο 45 λεπτά για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ που κάνετε μια απόπειρα να απαντήσετε στι ερωτήσει. Και τώρα έχω μια ολόκληρη παρουσίαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η Κομισιόν. Α, εδώ είστε. Συγγνώμη, Εμμανουέλ. Κοίτα, τι έκανα. Προσπαθούσα να σα αγνοήσω. Δεν τα κατάφερα. Εδώ είστε όμω. Συγγνώμη, λοιπόν. Απλώ μία εικόνα δώστε μα τη άλλη έκθεση. Και ζητώ συγγνώμη, βεβαίω. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο διότι από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει χρόνος και να απαντήσετε και στην ερώτηση της Κριστίν. Μήπως θέλετε να απαντήσω μόνο ή να κάνω και σύντομη παρασία. Αν μπορείτε να απαντήσετε στα σύντομα και στις δύο και δεν πειράζει και μετά ε, να αφιερώσετε τα υπόλοιπα λεφτά στην παρουσίασή σας. Για να απαντήσω λοιπόν απλώς ε, στις ερωτήσεις σας για το κράτος δικαίου. Πράγματι, ξεκίνησε η διαδικασία του άρθρου 7 για την κατάσταση στην Πολωνία και η ερώτησή σας είναι τι γίνεται με την κατάσταση στην Ουγγαρία. Και εδώ λοιπόν να σας πω ότι στην περίπτωση της Ουγγαρίας αυτό που κάνει είναι να παραβαίνει με κυρώσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα, ε, ε, διότι στην περίπτωση της Πολωνίας, να σας υπενθυμίσω ότι τα πρώτα θέματα τα οποία ετέθησαν αφορούσαν το συνταγματικό δικαστήριο, για παράδειγμα. Πρόκειται για ε, καταστάσεις δύσκολα μπορούμε να τιμωρήσουμε με κυρώσεις. Σε περίπτωση, στην περίπτωση της Ουγγαρίας, και κάτι, αυτό δεν είναι και πολύ συχνό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πολλές διαδικασίες επί παραβάση, συντονισμένα, Για παράδειγμα, ερωτήθηκε το δικαστήριο το Δεκέμβριο για την κοινωνία των πολιτών και για το νόμο για την ε, εκπαίδευση. Ε, προσφύγαμε στο δικαστήριο, το δικαστήριο εξετάζει το ζήτημα. Ε, όσον αφορά το άσυλο και την νομοθεσία για το ε, άσυλο, ξεκίνησε και μια αιτιολογημένη γνώμη για την ε, διαδικασία αυτή. Ε, στην περίπτωση της Πολωνίας δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε μέσω επιβολής κυρώσεων. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να χρησιμοποιεί τις κυρώσεις και να προσφεύγει στο δικαστήριο αν δεν έχει ρυθμιστεί το ζήτημα. Στην περίπτωση της Πολωνίας είχαμε μια μεταρρύθμιση του συνταγματικού συστήματος την οποία ακολούθησε και το σύνολο ε, της δικαιοσύνης. Επομένως, πρόκειται για διαφορετική κατάσταση. Όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, συμφωνώ απολύτως ε, στην παρουσίαση μου, την οποία δεν θα κάνω. Ένας από τους τομείς ε, στους οποίους υπήρξε πρόοδος το 2017 και είχαμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε την συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ακριβώς για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν ε, τη βία κατά των γυναικών. Ήταν πολύ σημαντική η όλη διαδικασία για να ξεκινήσει αυτή η δυναμική διαδικασία και φυσικά υπάρχουν και συγκεκριμένα θέματα και πιο συγκεκριμένα η ε, συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Και εδώ πρόκειται και για θεσμικά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να κυρώσουμε αυτή τη στιγμή ε, τη σύμβαση ε, το συντομότερο δυνατόν και τη συγκεκριμένη ερώτηση της τροποποίηση τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων για να συμπεριλάβουμε τα αναπορικαγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και αν ναι πώς. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για αναθεώρηση της χάρτας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σήμερα η πρόκληση για όλους εμάς ε, εδώ δεν είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε κανόνες, ε, αλλά ε, την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, δηλαδή η δυνατότητα επιβολής ε, των κανόνων της χάρτας και πραγματικά αυτή είναι η πρόκληση σήμερα και ο οργανισμός ε, μας βοηθά πάρα πολύ σε αυτό. Πρέπει να εφαρμόζει αυτό το δίκαιο, το υπάρχει εδώ και 10 χρόνια πλέον είναι δεσμευτική η χάρτα και ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τα δικαιώματα που προβλέπονται από το χάρτη σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό φυσικά μας αφορά όλους, διότι τα, οι κανόνες υπάρχουν, τα δικαιώματα υπάρχουν και το πραγματικό πρόβλημα είναι η αποτελεσματικότητά τους. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να σήξω στην παρουσίαση που δεν θα κάνω, είναι ότι το 2017 προχωρήσαμε, θέλω να πιστεύω, στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το χάρτη. Και φυσικά το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνία των πολιτών η οποία θα είναι ελεύθερη, δυναμική και ούτω καθεξής και φυσικά ένα από τα βασικά ερωτήματα το οποίο θα προκύψει και για σας τις επόμενες εβδομάδες είναι το νέο πολιτες πλαίσιο στο οποίο έχουμε δύο προγράμματα τα οποία θα είναι ουσιαστικά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, το πρόβλημα για τα δικαιώματα και τις αξίες και το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη. Το να έχουμε λοιπόν αποτελεσματικά δικαιώματα της χάρτας σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνία των πολιτών που έχει κίνητρα και που δραστηριοποιείται εξετάζουμε και τα θέματα τα οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο και ερχοζόμαστε ε, ενεργά για αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στις πτυχές της επίλυσης των διαφορών. Δεν ξέρω πώς τα λέμε στα γαλλικά και έχουμε την ε, δράσεις, τις στρατηγικές ε, και τις προσφυγές που χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Μπορούμε να βοηθήσουμε και υπάρχουν αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας για να αντιδράσουμε στον τομέα αυτό. Το να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και ε, διοικήσεις που λειτουργούν αποτελεσματικά. Έχουμε κάποια πράγματα που αφορούν το δίκτυο ε, των ε, κυδεμόνων παιδιών ε, σε περίπτωση μετανάστευσης. Έχουμε εφαρμόσει, μάλλον έχουμε συστήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την κυδαιμονία αυτών των παιδιών και την αναδοχή και ε, αυτό πιστεύουμε θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους και φυσικά χρειαζόμαστε και την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων της χάρτας το οποίο εξαρτάται και από τα εθνικά δικαστήρια. Ε, και πέραν της κατάστασης στην Ουγγαρία έχουμε εφαρμόσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και μια πολιτική η οποία στόχο έχει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ποιότητα της δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Ε, στο τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ε, ε, ψήφισμα για το scoreboard για τη δικαιοσύνη που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μανουέλ, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γιατί ε, θέλαμε να περιγράψεις και την ε, έκθεση και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν μετρήσαμε καλά τον χρόνο, 45 λεπτά για την έκθεση και τις ερωτήσεις ε, δεν αρκούσαν. Εγώ φταίω προσωπικά. Θα σας καλέσουμε ξανά για το θέμα αυτό και για να μιλήσουμε για τα θέματα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη γιατί η διερμηνία θα τελειώσει ακριβώς στο προβλεπόμενο ωράριο. Στις 6.30 ακριβώς. Οπότε να ευχαριστήσω τον Μάικλ Φλάχερτη και τον αγαπητό συνάδελφο πάρα πολύ και την ομάδα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να περάσω στο επόμενο θέμα τώρα κατευθείαν. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο 23. 45 λεπτά και για αυτό το θέμα. Όπως ξέρετε, Στις 17 Μαΐου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Στην παράγραφο 10 το Κοινοβούλιο έδωσε εντολή στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να ξεκινήσει διαδικασίε να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση. Όπως ξέρετε η κυρία Σαρτζεντίνη ορίστηκε συντάκτη στι 11 Ιουλίου πέρσι. 263 τροπολογίε υποβλήθηκαν. και η σημεία για τις τροπολογίες ήταν 15 Μαΐου. Έκτοτε ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές ε, προσπαθούσαν να καταλήξουν σε κάποια ε, συμφωνία επί των συμβαστικών τροπολογιών. Οπότε χωρίς άλλη καθυστερή θα δώσω αμέσως τον λόγο για την ανταλλαγή απόψεων επί των ε, τροπολογιών. Πρώτα απ' όλα βεβαίως στην εισηγήτρια για 10 λεπτά σας παρακαλώ η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ως εμείς ε, εργαζόμαστε στην ε, έκθεση αυτή, συνεδρίαζε σήμερα και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και ψήφισαν να αλλάξουν το Σύνταγμα και ένα νέο νόμο περί Μίκιο και πέρασαν και τα δύο. Και είναι νομίζω μια θλιβερή ημέρα την Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων είναι λυπηρό να βλέπουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίζει, να μειώσει την δυνατότητα των Ούγγρων να διευκολύνουν την ε, ευημερία των προσφύγων στην κοινωνία τους. Ε, υπό το φως αυτών των ψηφοφοριών θα ζητήσω από τους κοιοδησηγητές να κάνουν λίγη υπομονή γιατί θα θέλαμε βέβαια να ενημερώσουμε και τις συμβαστικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε την Δευτέρα να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρε και όπως ξέρετε εργαζόμαστε επί τη βάση ε, πηγών που τις έχουμε ελέγξει, της νομοθεσίας, ε, των αποφάσεων των δικαστηρίων, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έγκυρων πηγών Γι' αυτό μέχρι τώρα βλέπετε παραδείγματος χάρη την δυνατότητα που είχαμε να εργαστούμε με βάση τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Τώρα λοιπόν θα εργαστούμε με βάση την σημερινή ψηφοφορία. Και πάλι λοιπόν για την σημερινή ψηφοφορία η Επιτροπή αυτή πριν από λίγες εβδομάδες ζήτησε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο να καθυστερήσει η ψηφοφορία για τον νόμο περιμικιών μετά τα συμπεράσματα της Επιτροπής της Βενετίας. Νομίζω ήταν ένα λογικό αίτημα. και ζητούσαμε ακριβώ να υπάρξει σεβασμό στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν συνέβη και είναι πραγματικά κρίμα. Επί των συμβιβαστικών προτάσεων. Ε, επί των τροπολογιών. Πράγματι υπήρχαν 263 και τις τελευταίες ε, δύο εβδομάδες ε, προσπαθήσαμε να συμβάσουμε όσο δυνατόν περισσότερες και έχουμε γύρω στις 50 συμβιβαστικές από όλες τις ομάδες που υπέβαλαν τροπολογίες. Παραδείγματος χαρήν περιέλαβα σαφεστερή διατύπωση για την ανάγκη καταπολέμησης του αντισημιτισμού γιατί κάποιοι συνάδελφοι διακομματικά μου υπέβαλαν τέτοιες διατυπώσεις αυτό έχει περιληφθεί και προσπάθησα να δεχτώ και τροπολογίες από Ούγγρους συναδέλφους του ΕΛΚ γιατί πολλές από αυτές τις τροπολογίες είχαν ουσία δεν θέλω να χαθεί η δυνατότητα να διορθώσω τη διατύπωσή μας και τα γεγονότα οπότε έχουν περιληφθεί αυτά όμως κάποιοι από αυτούς τους συναδέλφους δεν θέλησαν να περιληφθούν στις συμβαστικές προτάσεις οπότε το κανονίσαμε αυτό αλλιώς έτσι ώστε να μην χαθεί η ουσία αλλά και οι άνθρωποι αυτοί να μην εμφανίζονται στην χώρα τους ότι είναι μέρος αυτού του συμβιβασμού. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πως αυτά είχα να πω τελικά αυτή τη στιγμή. Άκουσα τους ε, συναδέλφους, ε, αλλά έχω την εντύπωση πως οι σκιώδεις εισηγητές ε, θεωρούν ότι έχουν περιληφθεί όλα όσα ήθελαν. Α, και τέλος, τέλος, επέλεξα και ζήτησα το ίδιο και από τους συζητητές ε, να εργαστώ μόνο με βάση επίσημες πηγές και όχι Μίκιο. Και ήμουν ε, πολύ επίμονη σε αυτό. Οπότε οτιδήποτε αναφέρουμε είναι από διεθνείς οργανισμούς και όχι την κοινωνία των πολιτών και θέλω ε, να σας παρακαλέσω να γίνει αυτό και στις ε, χωριστές ψηφοφορίες για να είναι ευκολότερη η συζήτηση μετά, για να μην συζητάμε το εάν είχε προκατάληψη η πηγή ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Ακούστε με τώρα. 17.45 τελειώνουμε όπως και να έχει. Έχω πολλούς ομιλητές, δεν ε, θα πω τίποτα στους και ε, με έχουν ενημερώσει για τις αλλαγές. Μετά περνάμε στους ομιλητές που θα τελειώσει 17.45. Δεν θέλω παράπονα. 6.30 ώρα τελειώνουν ε, οι διερμηνείς. Παρακαλώ, Μαρή Κριστίν, λίγο σύντομα. Ναι, οι διερμηνείς, οι μας λένε στα ακουστικά ότι η διερμηνία θα συνεχιστεί μέχρι τις 6.30 ε, που είναι το ωράριό τους. Οπότε δεν ξέρω γιατί λέτε 17 και 45. Διερμηνή είναι εδώ μέχρι τι 6.30. Και ισχύει αυτό το οποίο λέει η κυρία Βεζιά. Ναι, ναι, για την ε, υπηρεσία των ε, ναρκωτικών πράγματι. Μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα ότι τελειώνει 5 και 45. Μάλιστα. Η κυρία Μετσόλα έχει αντικατασταθεί από τον κύριο Μπόνι για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μέτσολα ήταν έρθει αλλά είχε κάποιο, κάποια ανελημμένη υποχρέωση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτή η έκθεση, έκθεση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ομάδα μας. Το μεγαλύτερη πλειονότητα των ε, τροπολογιών είναι από μέλη του ΕΛΚ. Κάποιες πηγαίναν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με την ψηφοφορία της Δευτέρας στη Λίμπε, όλα τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για την έκθεση. Γι' αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των σκιωδών, επέμεινα να γίνουμε, ε, γίνουν ξεχωριστές ψηφοφορίες για πολλές ε, κρίσιμες τροπολογίες, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να εκφραστεί κατά συνείδηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την εισηγήτρια και τους υπολείπους σκιώδες που δέχτηκαν το αίτημά μου αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τώρα εγώ δεν ήμουν στον κατάλογο των ομιλητών κατά τα άλλα. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Ο πρόεδρο, όχι, όχι, δεν θα προλάβουμε. Δεν το ξέρω. Δεν μπορείτε να πάρετε δύο φορέ το λόγο, αλλά τώρα όσο. Πολύ σύντομα λοιπόν, κύριο Μπόνι, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ε, να διευκρινίσω ότι αυτό δεν στρέφεται κατά της Ουγγαρίας σαν χώρα, σαν λαό, σαν τους πολίτες της Ουγγαρίας. Ε, προσπαθούμε να πούμε ξεκάθαρα και με αυστηρότητα ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας παραβιάζει μια σειρά από κανόνες και η τελευταία της απόφαση η σημερινή για το νομοθετήμα που υποτίθεται ότι θα σταματήσει τον Σόρος ε, ψηφίστηκε σήμερα από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο χωρίς να ακούσουν, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της ε, Βενετίας. Μίλησα σήμερα με την Υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας και με, με υποσχέθηκε ότι θα το είχαν καθυστερήσει και θα είχαν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους και την Τροπή της Δεν το έκαναν. Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο το γεγονός ότι ποινικοποιούν τους άστεγους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα μέτρα τα οικονομικά που σκοπεύουν να πάρουν έναντι των προσφύγων και, τους μετανάστες, και των μεταναστών. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προ τον ουγγρικό λαό και προ την ουγγρική κοινωνία των πολιτών, ότι δεν είναι μόνοι του. Σα ευχαριστώ και ο Βάιντεν Χώσερ από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να φτάσουμε ω εδώ και να έχουμε την επόμενη Δευτέρα μια έτοιμη έκθεση και αυτό οφείλεται στο ότι τα επιχειρήματα πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά και βεβαίως ε, δεν ε, ε, είναι εύκολο κάτι τέτοιο όταν μιλάμε για τα συμπεράσματα αυτά. Πρέπει να πούμε ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ διαφανής, ανοιχτή. Ακούστηκαν όλα τα διαφορετικά επιχειρήματα από όλες τις σκοπιές. Θεωρώ ότι η προσέγγιση της εισηγήτριας ήταν πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή περιορίστηκε και βασίστηκε σε επίσημες πηγές μόνο, καμία εκτίμηση, καμία κρίση, αλλά μόνο βασίστηκε σε ε, επίσημα στοιχεία για την έκθεση αυτή. Είχαμε πολύ έντονες ε, συζητήσεις ε, με τους ηγητές. Ήταν ουσιαστική η ατμόσφαιρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ την εισηγήτρια για το ότι ε, ασχολήθηκε συστηματικά με το θέμα, περιέλαβε όλες τις απόψεις και προσπάθησε να περιλάβει όλα τα επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, σημεία κριτικής και νομίζω άρα ότι τελικά ε, έχουμε ένα καλό μήνυμα για το ότι ε, ο κοινοβουλευτισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζει ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το ECR, Μάρεκ Γιούρεκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα πολιτικό που διχάζει και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να βαθύνει την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενισχύσει τις συγκρούσεις. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι απολύτως ανεύθυνο αυτό που γίνεται και όχι μόνο ανεύθυνο. Είναι μια ηθελημένη προσπάθεια να καταδικαστούμε και οι χώρες μας οι δημοκρατικές που έχουν μια άλλη προσέγγιση να μην γίνουν σεβαστές. Και αυτό έρχεται αμέσως μετά το Brexit. Με εξέπληξε ολότε. Γιατί, Γιατί είπε ότι έχουμε... είπε μάλλον ότι η επίθεση αυτή που γίνεται στην Ουγγρική κυβέρνηση, στην Ουγγαρία, δεν είναι επίθεση προς τους Ούγγρους πολίτες. Αλλά ας καταλάβουμε λίγο τι κάνουμε εδώ. Οποιαδήποτε κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να κάνει τις δικές του επιλογές δημοκρατικά. Υπάρχει αντιπολίτευση στην Ουγγαρία. Μπορεί να μην συμφωνεί ο λαός με την ε, κυβέρνηση και τότε μπορεί να τους αλλάξει σε εκλογές. Όμως σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχει συνεργασία μέχρι να ακούσουμε όλες τις απόψεις όλων. Να είμαστε ανοιχτοί στις ε, διαφορετικές απόψεις. Ε, δεν Πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση η συγγήτρια μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ανοιχτή. Η συμπεριφορά έναντι των, ε, της Ουγγαρίας είναι απαράδεκτη. Αποτελεί ε, επίθεση κατά των δημοκρατικών διαδικασιών της Ουγγαρίας. Στο σημείο 7 ασκούμε κριτική επειδή άλλαξαν το σύνταγμά τους. Στο σημείο Καταδικάζουμε το γεγονός ότι η Ουγγρική ε, κυβέρνηση έκανε μια δημόσια διαβούλευση. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Ενωμένοι θα έπρεπε να ήμασταν εναντίον αυτής της έκθεσης, αυτού του εγγράφου, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει σε συνέπειες και για, τις σχέσεις και, για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και για τη σχέση της Ένωσης με την Ουγγαρία. Γιατί είναι σαν να λέμε ότι δεν μπορεί κανείς να έχει μια διαφορετική γνώμη. Σόφι από την πλευρά της Άλτε, καθιστώντας του Σκιώδη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Και θα ακολουθήσω την πρόταση της να μην υπάρξουν αναφορές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ως πηγές, αλλά θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε το μακρύ χέρι του Ορμπάν να μας υπαγορεύει τι είναι ε, πηγή αξιόπιστη και τι όχι. Θα του δώσουμε τέτοια δυνατότητα. Μην ανησυχείτε, θα ακολουθήσω την πρότασή της. Αλλά εδώ που προσπαθούμε να αναφερθούμε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να μην παραπέμπουμε σε αυτές γιατί αυτό φαίνεται σαν να, είναι, σαν τις ε, καθιστά ύποπτες. Ε, δεν αναφέρεται μόνο σε μη κυβερνητικέ οι οποίε μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον Σόρο, αλλά και από άλλε πηγέ. Αναρωτιέμαι, πόσα, πόσα κόμματα στην Ευρώπη, ορισμένα από τα οποία είναι μέλη του ECR, έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον κύριο Μπάνον και το κόμμα του κυρίου Ορμπάν έχει σχετικέ δωρεέ λάβει. Επομένω, την διαφάνεια που διακηρύττει για του άλλου, καλά θα κάνει να την εφαρμόσει και στην περίπτωση τη δική του. Σκιώδη για την Γκουε, κυρία Φρυχιάτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία κατάφερε με πολύ νυφάλιο τρόπο να διεξάγει αυτό το έργο. για να είμαι ειλικρινή, δεν θα είχα καταφέρει να <laughs> διατηρήσω την ψυχραιμία και την εφαλαιότητα που εκείνη κατάφερε να, ε, κρατήσει αν μου, στη θέση τη. Πρέπει να προχωρήσουμε και για να γίνει αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι τελείως άμεμπτη η έκθεσή μας. Και απαντώ και έτσι εμέσω στην ε, σοφή ε, την κυρία Τφέλτ, γιατί και εγώ απέσυρα κάποιες από τις ε, τροπολογίες μου, γιατί αν χρησιμοποιήσουμε μόνο τις επίσημες πηγές, αυτό δίνει τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι η έκθεσή μας είναι στέρεη και τελείως άμεμπτη. Ε, μία από τις κυριότερες κατηγορίες που μας προσάπτει το ΦΙΝΤΕΣ είναι ακριβώς αυτή. Έτσι λοιπόν, εάν δεν κάνουμε τι παραπομπέ τη κυβερνητική οργανώση κτλ., πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία σε ένα ζήτημα ευαίσθητο. Θα επαναλάβω και εγώ ότι η έκθεση αυτή δεν είναι μια έκθεση κατά τη Ουγγαρίας. Αυτό πρέπει να το επαναλάβουμε. Το να ασκεί κανείς κριτική σε μια κυβέρνηση δεν είναι κριτική σε μια χώρα. Αυτό ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις που έχουμε ασκήσει κριτική. Ε, είχα υποβάλει πολλές ε, τροπολογίες. Αλλά ε, συνεργάστηκα και συμμετέχω τώρα σε όλους τους συμβιβαστικές λύσεις. Όταν η, μια χώρα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συμφωνήσει να τηρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης, ανάμεσα στα οποία είναι μια σειρά κριτηρίων για το σεβασμό του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, σε όλες τις μορφές της. Η δημοκρατία δεν είναι το δίκαιο της πλειοψηφίας. Είναι επίσης και ο σεβασμός της μειοψηφίας. Δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε εκείνους που έχουν μια διαφορετική άποψη από την πλειοψηφία και να λέμε ότι αυτό είναι δημοκρατία. Δυστυχώς ε, το βλέπω αυτό να διαμορφώνεται ω τάση σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να το α, ε, σταματήσουμε. Καταδικάζω και εγώ το γεγονό ότι σήμερα υπερψηφίστηκε ο νόμο για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Ουγγαρία, χωρί να περιμένουν τη γνωμοδότηση τη ε, ε, Επιτροπή τη Βενετία. Ε, φέρνει πολύ προ τα πίσω την Ουγγαρία, προσπαθώντα να κάνει. να, να, να μπλέξει διαφορετικά πράγματα, όπω για παράδειγμα την ε, βοήθεια σε πρόσφυγε ή μετανάστες και την τρομοκρατία. Και αυτό πιστεύω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα και ακόμα πιο καταδικαστέο σήμερα την Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων. Σα ευχαριστώ. Η FDD δεν μας έχει, ούτε η ΕΝΕΦ δεν μας έχουν δηλώσει σκιώδη γιατί Επομένω, θα συνεχίσω με τον κατάλογο των ομιλητών. Δύο λεπτά, το μέγιστο ο καθένα παρακαλώ. Ο κύριος Λόπες Ογκυλάρ παρακαλώ, μέχρι δύο λεπτά. Λιγότερο θα χρειαστώ. Το ζήτημα είναι πολύ πολιτικό, είναι ουσιαστικά πολιτικό, αλλά το ερώτημά μου είναι τεχνικής φύσεως. Μετά τους ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, υπάρχει τίποτα στη διατύπωση που να προβλέπει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουμε επόμενες φάσεις της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να περάσουμε από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου, να πάμε σε αυτά που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο. Πρόεδρο, βεβαίω αυτή η συζήτηση βοηθάει να επιβάλλουμε ερωτήματα στην εισηγήτρια. Ευχαριστούμε κύριε Λόπε Αγγιλάρ. Και Γκαγκάλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. μαζί με τους συναδέλφους από το ΕΛΚ ε, από την Ουγγαρία υποβάλαμε 130 τροπολογίες που είναι περίπου το 50% όλων των τροπολογιών προς την έκθεση της κυρίας Αργεντίνη. Ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών ήταν για να δείξουμε ότι δεν υπάρχει ε, λόγος να υπάρξει διαδικασία άρθρου 7 και υπάρχουν και πάρα πολλά λάθη, παρανοήσεις ε, και σφάλματα και ε, φυσικά και προκατηλημένες πολιτικές απόψεις οι οποίες είναι παραπλανητικές. Αυτό το στόχο έχουν οι τροπολογίες μας. Η κυρία Σαρχεντίνη πήρε κάποιες προτάσεις από αυτές τις τροπολογίες ε, οι οποίες δεν βελτιώνουν το κείμενο στην ουσία στην πραγματικότητα απλώς αλλάζουν το κείμενό μας και δεν αλλάζουν δηλαδή ούτε καν τα λάθη όσον αφορά τα γεγονότα στο κείμενό της. Η απόφαση υπάρχει ήδη, είναι ηλυμένη και χρησιμοποίησε κάποιες από τις τροπολογίες απλώς ε, για να ε, τηρήσει τα προσχήματα, κάποια κομμάτια των τροπολογιών μας για να πει ότι έλαβε υπόψη τις τροπολογίες μας και δεν συμφωνούμε φυσικά με αυτό. Γι' αυτό και τη ζήτησα να μην συμπεριλάβει τις τροπολογίες μας στις συμβαστικές της ε, προτάσεις. Επίσης ε, θα πρέπει να σας πω ότι είδα τις συμβιβαστικές τροπολογίες και η έκθεση εξακολουθεί να αναφέρεται σε αρκετές περιπτώσεις ε, οι οποίες έχουν ήδη κλείσει από την Ουγγρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα. Τα κράτη-μέλη έχουν πλήρη αρμοδιότητα στα θέματα αυτά και δεν ε, επηρεάζουν αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες παρουσιάζονται ως μητέρες στα ουγγρικά σχολικά βιβλία. Είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Ε, εγώ είμαι περήφανη γι' αυτό. Ή για παράδειγμα η ελάχιστη σύνταξη. Αν δείτε τα στοιχεία, τα νέα κράτη-μέλη με την ιστορία τους. Αν δούμε το πολύ χαμηλό επίπεδο ελάχιστων ε, ε, συντάξεων θα μπορούσε να ξεκινήσει διαδικασία επιπαραβάση εναντίον όλων αυτών των χωρών. Νομίζω ότι είναι λίγο υπεροπτικό όλο αυτό και λίγο ε, υποκριτικό. Όσον αφορά τις διαδικασίες επί δεν νομίζω ότι η Ουγγαρία έχει χειρότερες επιβέωσεις από άλλες χώρες. Τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος δικαιοσύνης μας είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τις ε, ε, απόψεις κυρίας Αρχεντίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ναι, εγώ είμαι από την ίδια χώρα, αλλά έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Σαρχεντίνη έκανε μια πολύ ισορροπημένη ε, πρόταση ε, και γι' αυτό ακριβώ την ευχαριστώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ και τους κοιόδης συγητές. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν χρειάζεται τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό το οποίο συνέβη σήμερα το απόγευμα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Ε, η νομοθεσία που πέρασε νομίζω ότι αποδεικνύει ακόμα καλύτερα ότι ε, ανησυχεί τους πάντες ε, και Νομίζω ότι η Ουγγαρία δεν έχει δημοκρατία με ευρωπαϊκού όρου. Δημοκρατία δεν είναι η δικτατορία τη πλειοψηφία. Δημοκρατία σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη και τι απόψει των άλλων και ε, η ποικιλομορφία πρέπει να εκφράζεται και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι είναι απολύτω απαραίτητο για άλλη μια φορά να ε, ε, δούμε τα πράγματα όπως είναι. Πρόκειται για μια αντικειμενική έκθεση, το ανέφερε και ο κύριος Μπόνι. Πρόκειται για επικρίσεις προς την κυβέρνηση και στην παρούσα πολιτική ε, της και όχι κατά της Ουγγαρίας και των Ούγγρων. Και γιατί αυτό, διότι υπάρχει μια άλλη Ουγγαρία, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και εγώ είμαι περήφανος που εκπροσωπώ αυτή την άλλη Ουγγαρία. Αυτή την Ουγγαρία η οποία ε, σηκώνεται για να υπερασπίσει τα ευρωπαϊκά ε, κεκτημένα, τις ε, φιλελεύθερες αξίες ε, και δεν θέλει να έχει έναν αλεύθερο κράτος ε, κατά αυτής της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. E, Σα ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να συγχαρώ την εισηγητρία. Γιατί πιστεύω ότι κατέληξε σε συμβιβαστικές λύσεις που είναι πολύ καλά ισορροπημένες. Ήσασταν ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις κατά τη σύνταξη Τη έκθεση και την υποβολή των τροπολογιών. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ακροδεξιά να σηκώνει κεφάλι σε πάρα πολλές χώρες. Όμως, σε πολλές χώρες αυτή η έκθεση του λαϊκισμού εν μέρει οφείλεται στο ότι βλέπουν την Ουγγρική κυβέρνηση ως υπόδειγμα. Στην Ουγγαρία βλέπει κανείς ξεκάθαρα ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης παραβιάζουν το άρθρο 2 της συνθήκης. Η Ουγγρική κυβέρνηση διεξάγει μία εκστρατεία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα της και επιδιώκει να είναι όλο και περισσότερο πιο, πιο κοντά στη Ρωσία παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας μην ξεχνούμε ότι και η πολωνική κυβέρνηση εμπνέεται από αυτά που βλέπει να γίνονται στην Ουγγαρία και η Πολωνία θα αντιμετωπίσει τη διαδικασία του πρώτη παραγράφου του άρθρου 7 της συνθήκης. Θα έλεγα ότι είναι δίκαιο να έχουμε μια αντίστοιχη διαδικασία και για την Ουγγαρία. Η κυρία Γκόμες, σύντομα μόνο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές που κατέληξαν σε μια ισορροπημένη έκθεση και που περιγράφει, ε, μάλλον που, που, που αναλαμβάνουν, με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κυβέρνηση που έχουμε στην Ουγγαρία, η οποία έχει προχωρήσει σε ενέργειες που μας ντροπιάζουν όλους. Είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία. Και θα επαναλάβω, δεν είναι μια θέση κατά της Ουγγαρίας, κατά του λαού της Ουγγαρίας. Είναι μια θέση υπέρ εκείνων που συνεχίζουν να υπερασπίζονται τη δημοκρατία στην Ουγγαρία και συνεχίζουν να υπερασπίζονται το ευρωπαϊκό τρόπο ζωής απέναντι στους φασίστες και στο ολοκληρωτισμό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γιάροκα. με όρο του σεβασμό στη συνάδελφο κυρία Γκόμε. Θα διαφωνήσω μαζί τη, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την έκθεση τη κυρία Σαρτζεντίνη. Όλοι λέτε ότι δεν είναι κατά του λαού τη Ουγγαρία. Εάν δεν ήταν, δεν θα το θεωρούσαν δύο μέτρα και δύο σταθμά όλοι δεν θα προσπαθούσατε να υπερασπιστείτε τους, εκείνους που ασχολούνται με το τράφικινγκ στην Ουγγαρία σήμερα με τους λόγους σας, αλλά θα ήσασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό που γίνεται με την νέο νομοθεσία. με την έκθεσή σας κυρία Σαντζετίνη κάνετε, το κάνετε ακόμα πιο δύσκολο για τους Ευρωπαίους πολίτες να αντιληφθούν την κατάσταση στην Ουγγαρία και αποφασίσατε ότι οι τροπολογίε τις οποίες σας είχα υποβάλει δεν ήταν αρκετά σαφείς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεσή σας. Πιστεύω ότι δεν τολμήσατε να ακούσετε τις μη να, να, να μάλλον καταγράψετε τη θέση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην έκθεσή σας ακριβώς επειδή αυτοί οι θέσεις δεν είναι τεκμηριωμένες. Για αυτούς μιλούμε αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία, για οργανώσεις οι οποίες δεν είναι τεκμηριωμένες, δεν είναι επαγγελματικές, δεν εκπροσωπούν το λαό, δεν εκπροσωπούν την τοπική κοινωνία. Σας ζητώ λοιπόν να επανεξετάσετε το εάν θέλετε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, σα ζητώ να καταψηφίσετε ουσιαστικά την έκθεση την επόμενη Δευτέρα. Περνάμε στα υπόλοιπα μέλη και ο Ζάνιεφ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω στο σκέλος της συζήτησης που αφορά στη δημοκρατία, στην έννοια της δημοκρατίας. Επί 8 χρόνια ένας πακτολός χρημάτων έχει χρησιμοποιηθεί για να γίνει πλήση εγκεφάλου στους Ούγγρους πολίτες. Ούτε καν οι βασικές αρχές της δημοκρατίας δεν έχουν επιβιώσει στην Ουγγαρία από αυτή την κυβέρνηση. Έχει τόσο πολύ χρησιμοποιήσει τον έλεγχο της επί του τύπου η Ουγγρική κυβέρνηση που οι Ούγγροι πολίτες δεν μπορούν πια να έχουν ε, ασφαλή και σωστή πληροφόρηση. Είναι και ένας από τους λόγους που επανεξελέγει ο κύριος Ορμπάν με τέτοια μεγάλη πλειοψηφία. Νομίζω πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Πρέπει η Ευρώπη να επιδείξει αλληλεγγύη με εμάς, τους Ούγγρους. Μετά, για το λεγόμενο πακέτο νομοθετικών μέτρων για να σταματήσουν τους όρους. Να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχει καμία σχέση αυτή η νομοθεσία με το να σταματήσει την επιρροή του κυρίου Σόρος. Ο στόχος είναι να καπηλευτεί το φόβο η κυβέρνηση, το φόβο που δημιούργησε και να τον χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία, ως άλοθη, για να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης στην Ουγγαρία. Να χρησιμοποιήσει τα όργανα του κράτους με τρόπο που θυμίζει τις πιο μαύρες ε, σελίδες της, της ιστορίας της χώρας μου. Ε, υποστηρίζω πλήρως την έκθεση της κυρίας Αργεντίνη. Ευχαριστούμε κύριο Ζάερ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι μέλος ε, της Επιτροπής Λίμπη, αλλά έχω υποβάλει αρκετές ε, τροπολογίες. Η έκθεση της Επιτροπής σας είναι κατ' ουσίαν ένα κατηγορητήριο που βασίζεται σε αναλήθειες και ψέματα. Και έχουμε αυτήν την ταινία «Ο μάρτυρας» του Πίτερ Μπρούτσο. Μια σατυρική ταινία για τον ε, παραλογισμό του σταλινισμού. Και σε μια σκηνή αυτής της ε, ταινίας ε, ο δικαστικός κλητήρας μπλέκει το κατηγορητήριο με την τελική απόφαση η οποία έχει ήδη εκδοθεί. Και αυτό κάνετε και εσείς τώρα. Είστε και εισαγγελέα και δικαστής. Κατηγορείτε την ομπρική κυβέρνηση και τον ομπρικό λαό. Το ελάχιστο θα ήταν να μας δώσετε την δυνατότητα να υπερασπιστούμε εαυτούς. Ακούσαμε αναφορές ε, ε, που μιλάνε για αντικειμενικότητα σε αυτήν την συζήτηση. Δέκα ομιλητές ήταν κατά της Ουγγαρίας, τρεις υπέρ της Ουγγαρίας. 22 λεπτά οι ομιλητές κατά της Ουγγαρίας, 8 λεπτά για να απαντήσουν ε, οι ομιλητές υπέρ της Ουγγαρίας. Είναι δίκαιο αυτό στην δική σας την ε, χώρα κύριε Πρόεδρε. Και δεν είναι μόνο η διαδικασία με την οποία έχω πρόβλημα, αλλά και βεβαίως η ουσία της έκτασης, οι τροπολογίες μας. Γιατί αναφέρεστε σε κάθε δεύτερη πρόταση στο κράτος δικαίου. Κράτος ε, δικαίου σημαίνει ότι η συμπεριφορά των πολιτών ε, δεν είναι αυθαίρετη αλλά καθορίζεται από τον νόμο και το ίδιο ισχύει και για τη ΛΥΜΠΕ. Πρέπει να εργαστείτε εντός του πλαισίου των συνθήκων. και βεβαίως ε, έχετε πράγματα ασχετά με χαμηλές συντάξεις ή το ε, γεγονός ότι ένας εκδότης έκλεισε μια εφημερίδα ή υπάρχουν λίγες γυναίκες ε, στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Μα αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ενώ μιλάτε για αυτήν την ιδέα του κράτους δικαίου, είστε εξίσου αυθαίρετοι όσο και οι χειρότεροι δικτάτορες και λυπούμε που άκουσα τόσους πολλούς Πολωνούς ε, να μιλούν κατά της Ουγγαρίας. Ο πρόεδρος, δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ε, σοβαρά τώρα, τι, τι είναι αυτές. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Είναι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι όσοι ήθελαν τον λόγο μίλησαν. Δεν έχει απομείνει κανείς. Ε, δεν το μετράμε μαθηματικά ποιο μιλάει. Αν θέλετε περισσότερα άτομα με την άποψή σας να μιλήσουν, να έρθουν να μιλήσουν αν υπάρχουν στο Κοινοβούλιο. Και θα του αφήσουμε βεβαίω γιατί είμαστε δημοκρατικοί σε αυτή την Επιτροπή. Κύριε Γιούρεκ, όχι, όχι. Μην προσπαθείτε καν. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην εισηγήτρια, στην εισηγήτρια για να συνοψίσει. Κοιτάξτε, μην, μην ξεκινήσω τώρα. η κυρία Σατζεντίνη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έγιναν κάποιες ερωτήσεις ε, και θα απαντήσω. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ ε, ρώτησε το εάν υπάρχει στο ψήφισμα μετά από τις συμβαστικές προτάσεις η δυνατότητα να περάσουμε από το άρθρο 7 εδάφιο 1 στο εδάφιο 2. Η απάντηση είναι όχι γιατί το κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και να πω πως θα πρέπει να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, κατά το οποίο σημαίνει πλειοψηφία 2 τρίτων, οπότε Ας ε, ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτό. Και τι κάνουμε. Ουσιαστικά βάζουμε αυτό το ζήτημα ενώπιον του Συμβουλίου για να ντραπούν που δεν έχουν κάνει τίποτα τόσα χρόνια. Ε, ζητώ συγγνώμη λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κοιτάξτε, να απορώ λίγο, αλλά θα το βρω μετά γιατί εγώ διευκόλυνα την κυρία Γιουρόκα γιατί δεν ήθελε να εμφανιστεί στον κατάλογο ψηφοφοριών γιατί αυτό θα την έφερνε σε δύσκολη θέση στην χώρα της αλλά τώρα λέει πως έχει αποσύρει. Ο, εντάξει, έχω πρόβλημα, αλλά δώστε μου το γραπτός για να σβήσω το όνομά σας. Και θα βγάλω αυτά που αναφέρθηκαν. Μετά η κυρία Γκάλα, την οποία επίσης διευκόλυνα με τον ίδιο τρόπο. Εάν υποβάλλετε τροπολογίες 113 ε, ε, που έχουν κάποιο περιεχόμενο, ε, δεν μπορεί να λέτε πως μετά πρέπει να γνωρίσουμε αυτό το περιεχόμενο. Ξεκινήστε να δουλεύετε μαζί μας, σας διευκόλυνα εντός του συστήματος και το ίδιο έκανα και με άλλους. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να μιλήσετε με την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα εάν δεν σας αρέσει η διατύπωση για την θέση των γυναικών στην ουγγρική κοινωνία. Γιατί εγώ διευκόλυνα την κυρία Κουντρίτσα εδώ. Τέλος. Νομίζω πως υπάρχει κάποια παρεξήγηση με κάποιους ε, Ούγγρους ε, συναδέλφους ε, για την έκθεση αυτή. Το έχω ξαναπεί, είναι σαφώς μέσα στο ψήφισμα. Εμείς πήραμε την ανακοίνωση τη Κομισιόν το 2003 που κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε που ξεκαθαρίζει ότι ε, κοιτάμε πέρα από το ευρωπαϊκό και και την Νομοσία της Ένωσης. Γι' αυτό κάθε φορά που υπάρχει ένα κείμενο που λέει ε, αυτά δεν είναι δουλειά σας, ε, αυτό δεν ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αναμένω την ψηφοφορία τη Δευτέρα. Okay, thank you very much. Um, okay, that's the end of the debate. Um, thank you very... Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χειροκροτάτε κύριε Γιούρ. Είναι διαδικαστικό το θέμα σας. Αν είναι διαδικαστικό να σας ακούσω. Είναι διαδικαστικό. Ναι. Άρθρο 11 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άρθρο 11 διευκρινίζει σαφέστατα ότι οι ευρωβουλευτές πρέπει να σέβονται ένα τον άλλον και σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση, ακόμα και στην Επιτροπή μας, κανένας ε, δεν θα πρέπει να λέει ξενοφοβικά πράγματα και ε, πράγματα τα οποία είναι ασεβή. Ε, και δεν υπήρχε καμία ε, δήλωση σαν αυτά που είπε η κυρία ε, Γκόμες. Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε εδώ σήμερα είναι φρικτά. Δεν μπορεί να λέτε ότι συμπεριφορόμαστε σαν φασίστες. Νομίζω ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αντιδράσει, διότι είναι πάρα πολύ αυστηρά αυτά τα οποία ακούστηκαν και ναι, ήταν διαδικαστικό αυτό και θα ήθελα όλοι να σεβαστείτε το άρθρο 11 ε, στη διάρκεια της συνεδρίας Επιτροπής τα διαδικαστικά θέματα είναι θέμα λάθος χρονισμού. Η κυρία Γκόμης το είπε εδώ πριν από αρκετή ώρα, αλλά η παρέμβασή σας ε, ήρθε στην πιο δραματική στιγμή όταν ε, επέκρινε κάποιο άλλο μέλος γιατί επέκρινε την Επιτροπή. Να σας πω το εξή ότι πραγματικά διαλέγετε την κατάλληλη στιγμή. Αν θέλετε να κάνετε κάτι διαδικαστικό κατά της κυρίας Γκόμης έπρεπε να το έχετε πει εκείνη τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περάσει ε, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν μπορούμε, ε, ενώ φεύγουν οι συνάδελφοι για το σημείο αυτό, να συζητήσουμε το θέμα. Άκουσα τι είπατε, ήταν πολύ έντονη συζήτηση και αυτό το οποίο δεν δέχομαι, πρέπει και εγώ πιστεύω να σεβόμαστε στον άλλον, ε, δεν ναι, σέβομαι, δεν δέχομαι αυτό που είπε και το μέλος ε, που δεν είναι μέλος της Επιτροπής ε, Λίμπε και ήρθε να μιλήσει ότι ε, δίνουμε το λόγο σε όλους, σε καμία περίπτωση δεν ακούσαμε την άποψη ολωνών. είμαστε πάντα δίκαιοι. Ευχαριστώ λοιπόν για την πειθαρχία σας και ευχαριστώ και για τα σχόλια. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Και έχουμε εδώ το διευθυντή, ο οποίος έρχεται στο βήμα. Αν μένετε για το σημείο αυτό, αν μένει οποιοδήποτε από εσά για το σημείο αυτό, σας παρακαλώ ε, ε, καθίστε στις θέσεις σας και οι υπόλοιποι αποχωρήστε ησύχως. Ε, Κάθε φορά που έρχεται ο διευθυντής ε, του κέντρου ναρκωτικών, προσπαθώ να σεβαστώ τα όσα κάνει ο οργανισμός σας. Παρακαλώ λοιπόν, όσοι θέλετε να παραμείνετε, παρακαλώ καθίστε. Αν θέλετε να συζητήσετε απλώς σας, παρακαλώ εκτός εθούσης. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο για σήμερα. Δόξα το Θεώ, γιατί ήταν μεγάλη μέρα. Η έκθεση αυτή λοιπόν δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουνίου και παρουσιάζει μια γενική εικόνα της κατάστασης των ναρκωτικών στα 28 κράτη-μέλη στην Τουρκία και στην Νορβηγία τα ε, στατιστικό δελτίο και οι 30 εκθέσεις αναχώρα συμπληρώνουν την έκθεση και υπάρχουν αντίγραφα εδώ στην αίθουσα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον ε, Διευθυντή του Κέντρου για μια σύντομη παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στα μέλη που θέλουν να ε, σχολιάσουν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τομέας πολιτικής και πολύ συχνά ε, δεν σας δίνουμε αρκετό χρόνο, δεν προβάλλετε αρκετά και δεν ε, προβάλλετε και το πόσο πολιτικά σημαντικό είναι το θέμα, αλλά δεδομένου των δραματικών συνεπειών και τη συζήτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, των ναρκωτικών στην κοινωνία μας είναι πάντα ε, λίγο το ενδιαφέρον που δείχνουμε. Σας το λέω αυτό εισαγωγικά και με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι εξελίξεις έχουμε από την τελευταία έκθεση που μας υποβάλλεται που ήταν πρόσφατη σχετικά. Κύριε Διευθυντά, έχετε λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Είναι χαρά και τιμή να έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάζω αυτή την επισκόπηση της κατάστασης των ναρκωτικών όπως παρουσιάζει και όταν ξεκίνησε η τελευταία εκδοχή της ε, έκθεσης ε, για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως ε, είπε και ο Πρόεδρος έχετε λάβει τις αναλυτικές πληροφορίες οπόμενο θα σταθώ στα ουσιαστικά της έκθεσης και θα σας κάνω και μια σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων που αφορούν την σε επιδόσεις του κέντρου αν μπορούμε να δούμε εδώ την επόμενη διαφάνεια. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι όπως αναφέρουμε και στην έκθεση υπάρχει αυξημένη διαθεσιμότητα και ε, πιο αγνή ε, παρουσία κοκαίνης. Ε, και πρέπει να το αναφέρουμε. Η κοκαίνη που πωλείται στην Ευρώπη έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα καθαρότητα τα τελευταία 20 χρόνια τα ε, μοντέλα χρήσης δεν είναι και τόσο σαφή, αλλά στην ανάλυση καταλήπων κοκαίνης ε, του νερού βλέπουμε ότι είχαμε αύξηση ε, σε 26 από τις 31 πόλεις αλλά η εικόνα είναι ανάμεικτη από τα στοιχεία που έχουμε και κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι ε, στα επίγοντα των νοσοκομείων ε, από τα στοιχεία που έχουμε η κοκαίνη είναι το δεύτερο ναρκωτικό το οποίο ανοιχνεύεται μεταξύ όσων φτάνουν ε, στα επίγοντα και σε ορισμένες χώρες μέλη όπως σε κάποιες, και σε κάποιες πόλεις όπως σε μια πρόσφατη μελέτη που διάβασα από το Λονδίνο διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ενδείξεις και σε άλλες μελέτες ότι υπάρχει αύξηση στη χρήση της κοκαίνης. Τώρα, ε, κατά πόσον η αύξηση αυτή ε, μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη ανάγκη θεραπείας δεν είναι σαφής ακόμα η εικόνα, αλλά αυτός είναι ένας από τους λόγους ε, ε που εξηγεί ότι κάποιος που χρησιμοποιεί ηρωίνη ε, μέχρι να φτάσει κάποιος ε, στο πρώτο αίτημα για θεραπεία είναι 8 χρόνια αφού ξεκινήσει την ε, χρήση. Και για αυτούς οι οποίοι είναι πιο κοινωνικά ενταγμένοι και χρησιμοποιούν κοκαίνη μπορεί να είναι αντίστοιχο το χρονικό διάστημα. Δεν εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι τα στοιχεία για τις αιτήσει για θεραπεία δεν αντανακλούν ακόμα την ίδια αύξηση που παρατηρούμε. Βλέπουμε όμω αύξηση στον αριθμό των ε, ε κρίσεων, των επιλεπτικών κρίσεων, ε, στις ποιότητε. Ε, ε, επίσης και έχουμε και κατασχέσεις. Στο Βέλγιο είχαμε τις περισσότερες κατασχέσεις και αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είχαμε στην Ισπανία τις περισσότερες κατασχέσεις. Ε, στην επόμενη διαφάνεια τώρα. Έχουμε και ανησυχίες για την παραγωγή ναρκωτικών στην Ευρώπη. Και εδώ η εικόνα και πάλι αλλάζει κάθε χρόνο. Αυτό το οποίο είναι γνωστό ήδη είναι ότι η Ευρώπη έχει γίνει σαφής και πολύ ισχυρός ε, ε παραγωγός MDMA, έκσταση, και ε, με τη Europol διαπιστώσαμε ότι αυξήθηκαν και τα εργαστήρια παραγωγής τα τελευταία χρόνια. Το έκσταση δεν παράγεται όμως για την ευρωπαϊκή αγορά μόνο, ε, γίνεται εξαγωγή και στις Ηνωμένε Πολιτείες και σε όλες ε, τις περιοχές του κόσμου. Και επίσης υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, δεν ξέρουμε τι σημαίνει, ότι τα τελευταία στάδια επεξεργασίας κοκαίνης και ηρωίνης γίνονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε ε, κατάσχεση ε, ε, σε κάποια εργαστήρια στην Ευρώπη όπου υπήρχε μορφήνη για ε, μετατροπή σε ηρωίνη και ε, ε, βάση για μετατροπή σε κοκαίνη και φυσικά αυτό το παρακολουθούμε με τη Europol. Φαίνεται ότι όπως αυξάνεται η πίεση για την ε, διαθεσιμότητα των χημικών πρόδρομων ουσιών και επομένως η αγορά προσπαθεί να διαφοροποιήσει την πρόσβαση σε αυτές τις ουσίες και προσπαθεί να προ... παράξει το προϊόν από τα χημικά τα οποία παράγονται για αυτούς τους σκοπούς όπως γίνεται στην αγορά της Ευρώπης. Είδαμε και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είχαμε εργαστήρια στα οποία παράγονται νέες ψυχοτρόπες ουσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ συνήθως αυτές οι ουσίες ε, ε, παλιά ερχόντουσαν από την Κίνα και όπως γνωρίζετε υπάρχει και σημαντική παραγωγή κάναβης στην Ευρώπη που χαρακτηρίζεται επίσης και από υψηλή συγκέντρωση και υψηλή ισχύ. Ε, Μιλώντα για την κάναβη, σας ευχαριστώ και μου αλλάξατε τη διαφάνεια, είναι το πιο ευρώ διαδεδομένο ναρκωτικό στην Ευρώπη. Αυξάνεται ο αριθμός ε, της ζήτησης ε, για θεραπεία και τα πρώτα αιτήματα για θεραπεία. Υπάρχουν μεγάλες καινοτομίες στις μορφές, τα προϊόντα και τα συστήματα παράδοσης και εδώ βεβαίως είναι πολύ σωστό να αναφέρουμε και τις αλλαγές που έχουμε και στις παγκόσμιες εξελίξεις. Θα ακούσατε ίσως για παράδειγμα ότι την περασμένη και την αυτή την εβδομάδα το, η Γερουσία και το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέα νομοθεσία για την ε, νομιμοποίηση της χρήσης κάναβης. Ε, υπάρχουν κάποιες πολιτείες στις Πολιτείες που έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο ή αποφάσισαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη ε, και στην Ελβετία γίνεται συζήτηση για κάναβη με λιγότερο από 0,8% THC, της ψυχοτρόπου ουσίας δηλαδή, ε, πωλείται νόμιμα στη χώρα και επίσης υπάρχει και η εξέλιξη των συνεπειών της εφαρμογής ε, της κυβερνητικής συμφωνίας στις κάτω χώρες. Ε, υπάρχει μια πιλωτική μελέτη η οποία καταρτίζεται για την ε, παραγωγή κάναβης ε, για τα coffee shops όπως είναι γνωστά ε, γιατί αυτό είναι και η πίσω πόρτα του συστήματος ανοχής των ναρκωτικών. Πολλά πράγματα συμβαίνουν κυρίως εκτός Ευρώπης τα οποία όμως σίγουρα θα έχουν μέσω μακροπρόθεσμα και συνέπειες για την κατάσταση των ναρκωτικών εδώ. Και βεβαίω υπάρχει και διασταύρωση αυτών των θεμάτων της κάναβη και της νομοθεσίας για την κάναβη με άλλα ε, ε, στοιχεία όπως για παράδειγμα οδήγηση και ναρκωτικά και είχαμε σχετική μελέτη για το θέμα αυτό την περασμένη εβδομάδα. Τώρα όσον αφορά τι νέε ψυχοτρόπες ουσίες, 51 ε, νέες ουσίες ε, διαπιστώθηκαν το 2017, περίπου 350 ουσίες ε, καταγράφονται ετησίω, δηλαδή βρήκαμε 350 από αυτές τι ουσίε κάπου στι ευρωπαϊκέ αγορέ πέρσι, αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε συνολικά 670 από αυτές τι ουσίε, οι οποίες ελέγχονται μέσω του Ευρωπαϊκού συστήματο Συστήματος Προειδοποίηση ε, για τα Ναρκωτικά, έχουμε μία μείωση σε σχέση με την ε, ε, μέγιστη τιμή που είχαμε το 2014 Έχουμε 101 την εβδομάδα, αλλά υπάρχουν περισσότερα περιστατικά θανάτων και οξείας ε, δηλητηρίαση, καθώς επίσης και αύξηση ε, της των ε, φαινοτανίνων που είναι κάποια συνθετικά οπιοειδή, τα οποία δημιούργησαν πολύ σημαντικά προβλήματα πρόσφατα και στις Ηνωμένε Πολιτείε οι ψυχοτρόπες ουσίες γίνονται πρόβλημα σε κάποιες χώρες ε, στα σοφρονιστικά καταστήματα, ιδιαίτερα τα συνθετικά καναβοηδή. Ε, έχουν διαπιστωθεί η παρουσία τους σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια δεν ε, υπάρχει παρουσία τους αλλού ακόμα. Υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα, θάνατη οξία δηλητηρίαση, αλλά και περιπτώσεις εκφοβισμού και έναρξη χρήσης στη φυλακή. Και βεβαίω ένα από τα προβλήματα είναι ε, η δυσκολία του σοφρονιστικού συστήματος να ανοιχνεύσει αυτέ τι ουσίες, γιατί για παράδειγμα μπορεί να τις ε, ψεκάσει κάποιο σε ένα χαρτί ή σε ένα ε, κομμάτι ύφασμα και μετά να περάσει παράνομα στη φυλακή. Ε, θα ήθελα να τονίσω, παρά το γεγονό ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε λεπτομέρειε ακόμα, ότι οι φυλακέ είναι πολύ σημαντικός ε, χώρος για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων των ναρκωτικών και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλο τμήμα των προβλημάτων και υπερβολική δόση είναι από χρήστε οι οποίοι ε, βγαίνουν από τη φυλακή και ξεκινούν ε, χρήση ναρκωτικών ε, με ίδιες ποσότητες ή ψηλότερες από ό,τι προηγουμένως και φυσικά μπορεί να υπάρξει υπερβολική δόση σε περίπτωση οπιοειδών. Εδώ τώρα στην επόμενη διαφάνεια αναφερόμαστε στη μείωση των περιστατικών υπερβολικής δόσης. Ε, τα σχετικά καλά νέα είναι ότι το 2016 είχαμε 9.000 θανάτους από υπερβολική δόση και λέω σχετικά καλά διότι πρέπει να το συγκρίνουμε και με την κατάσταση στις ΗΠΑ, Πολιτείες, όπου την ίδια χρονιά είχαμε 66.000 θανάτους από υπερβολική δόση και η μισή εξ αυτών ε, είχαν άμεση ή έμεση σχέση με φεντανίλ κυρίως σχετίζονται με ηρωίνη και άλλα οπιοειδή στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει σχέση και με συνθετικά οπιοειδή, αναφέρομαι στο φεντανίλ, αλλά υπάρχουν και φάρμακα και νομίζω ότι μία από τις βασικές προκλήσεις για μας ε, και είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θετικέ θετικές εξελίξεις σε κάποια κράτη-μέλη, ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες ε, και επενδύσεις ε, για τη χρήση του αντιδότου ναλοξών των οπιοειδών και μια και είμαστε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα ήθελα να τονίσω ότι μαζί με τη Europol έχουμε ασχοληθεί ε, με θέματα ε, επιβολής του νόμου και δημόσιας προειδοποίησης, διότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει οξία δηλητηρίαση, ακόμα και όταν έρθει κάποιος σε επαφή με αυτές τις ουσίες, όπως για παράδειγμα το φεντανίλ, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ολοκληρώσω με κάποια στοιχεία, αν μπορείτε να μου δείξετε την επόμενη διαφάνεια, Προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας του 2025 και όπως ξέρετε υπάρχει σαφής διέσμευση για περισσότερες υπηρεσίες με καλύτερη αξία. Φέτος λοιπόν είχαμε 64 ε, επιστημονικές δημοσιεύσεις 20 ε, συμβολές επιστομινικά άρθρα ή σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων για τα ναρκωτικά. Είχαμε επίσης 30 ε, εθνικές εκθέσεις ε, για ναρκωτικά που είναι νέα προϊόντα που περιγράφουν όχι απλώς την κατάσταση σε κάθε χώρα αλλά ε, θέτουν και την κατάσταση στη χώρα ε, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κατάστασης και είχαμε και τρεις βασικές δημοσιεύσεις φέτος, ε, την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά, αλλά επίσης και τον Ευρωπαϊκό Οδηγό για Κοινωνικές και Οικονομικές Απαντήσεις και αργότερα εντός του 2017 είχαμε και την έκθεση για τα ναρκωτικά στο Darknet, την οποία ξεκινήσαμε με τον Επίτροπο ε, Αβραμόπουλο στη Λισαβόνα και αν θυμάστε ε, πέρσι ε, ήμασταν στο δίκτυο των υπηρεσιών και οργανισμών δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και προεδρεύομαι. Τώρα, όσον αφορά την προβολή, είχαμε πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας. Είχαμε και νέα βίντεο και μικρά και μεγαλύτερα, τα οποία ε, κατέβασαν οι πολίτες 190.000 ε, φορές και 49 ψηφιακές εκστρατείες. Τώρα, οι υπηρεσίες ε, σε πολιτική έχουμε συμβάλει άμεσα σε 53 βασικές εκδηλώσεις ε, πέρσι και είχαμε πάνω από 300 συμβολές σε επιστημονική υποστήριξη, σε πολιτική και πρακτικές. Φτάνουμε προς το τέλος. Η υπηρεσία μας στην πράξη. Έχουμε βοηθήσει πάνω από 100 επαγγελματίες που ασχολούνται στον τομέα της ε, μείωσης ε, και παρακολούθησης ε, της χρήση ναρκωτικών και πάνω από 300 αξιωματικού υπαλλήλου μαζί με τη ΣΥΠΟΛ εκπαιδεύτηκαν και οργανίσαμε και την πέμπτη έκδοση ε, του Ευρωπαϊκού Θερινού Σχολείου για τα Ναρκωτικά με 51 ε, φοιτητέ ε, από 25 χώρες. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, απόδοση και μετά τα οικονομικά, οι επιδόσεις μας αυξήθηκαν και μπορέσαμε να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας, ιδίως στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας μας. Εφαρμόσαμε 97% των δραστηριοτήτων προτεραιότητας Ελένα, που σημαίνει δέσμευση να παρακολουθήσουμε να δώσουμε 100%. Βελτιώσαμε την ε, ε, ε επίδοση των πρωτορετήτων L2 στο 95% και για το L3 φτάσαμε στο 67% που είναι ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα που είχαμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Επίσης, εφαρμόσαμε τις αλλαγές στον οργανωτικό σχεδιασμό της υπηρεσίας μετά από την έγκριση της στρατηγικής και δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα δημόσιας υγείας. Όσον αφορά τα χρήματα τώρα, μία ερώτηση προς εσάς πριν τελειώσουμε. 37. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θα ρωτήσω τον κάθε ένα από εσά να ε, μου πείτε τι είναι, δεν θα το βρείτε ούτως ή άλλως. 37 cent ε, ε, δεν ε, ξοδεύει από τον προπολογισμό του το MCDD για το 2017. Είναι η καλύτερη επίδοση που είχαμε ποτέ και είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που καταφέρνουμε να έχουμε 100% των δεσμεύσεών μας για την εκτέλεση του προπολογισμού. Έχουμε όμως και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με την εκτέλεση των πληρωμών 94,7% και ε, τις δραστηριότητες οι οποίες μεταφέρονται, οι λεγόμενες ε, C8, εδώ έχουμε 94,6%, Φτάσαμε λοιπόν ε, σε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ακύρωσης ε, δεσμεύσεων, ε, και υποχρεώσεων και νομίζω ότι με αυτό το τελευταίο στοιχείο μπορώ να σας δείξω πολύ συγκεκριμένα όχι μόνο τι παραδίδουμε και τι πληροφορίες δίνουμε αλλά έχετε και ένα ακόμα παράδειγμα με την έκθεση που σας παρουσίασα σήμερα αλλά βλέπετε και ότι ο οργανισμός στηρεί τις δεσμεύσεις του να διατηρήσει και να βελτιώσει την παραγωγικότητα, τη λογοδοσία και τις επιδόσεις του. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στα μέλη. Ο εισηγητής μας για πολλές από τις ε, ψυχοτρόπες ε, ουσίες θα ξεκινήσει την συζήτηση. Ο κύριος Μπόνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο ε, Γκούτσιλ για την εξαιρετική του παρουσίαση και τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο μας μετέδωσε πληροφορίες, αλλά επίσης και για το τελευταίο σκέλος της παρουσίας της του, με το οποίο μας έδειξε την αποτελεσματικότητα της, ε, του οργανισμού του. Είναι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι προφανές ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την, τα προγράμματα για την πρόληψη και τη θεραπεία ε, της τοξικομανίας ταυτόχρονα με την παρακολούθηση της αγοράς βλέπουμε ότι η αν και τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα των ψυχοτρόπων ουσιών βελτιώνονται, μία από τις σημαντικές προκλήσεις που παραμένει είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η ζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό το διαπιστώσαμε ιδίω όταν μιλήσατε για τα ευρωπαϊκά εργαστήρια που παράγουν τέτοιες ουσίες εργαστήρια στην Ευρώπη. Και αυτές Εάν γνωρίζαμε καλύτερα πώς λειτουργούσε η αγορά, αν θέλετε, θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε την εξέλιξη στον χώρο των ψυχοτρόπων ουσιών. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει στην περίπτωση της χρήσης παραποιημένων ε, φαρμάκων ή της χρήσης τους εκτότης της συνταγογράφησης. Ε, θα ήθελα να μου πείτε για αυτό το θέμα. Τι κάνετε και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κυκλοφορία τους. Ναι, τη, την κυκλοφορία φαρμάκων χωρίς άδεια. Επίσης, πώς μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της ε, κυκλοφορίας. Ε, αναφέρετε κάποια εργαλεία, όμως την έκθεση σας λέτε ότι αυτά δεν είναι επαρκή για να παρακολουθούμε τις σημαντικές αλλαγές που σημειώνονται στην ε, χρήση των ναρκωτικών. για παράδειγμα, ότι θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες έτσι ώστε να γνωρίζουμε ε, τις αλλαγές ε, στο, μοτίβο της χρήσης κατά την άποψή σας. Τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να αναπτύξουμε αυτά τα νέα εργαλεία παρακολούθησης για να γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει με τη ζήτηση και με την κατανομή της ζήτησης, το είδος των ψυχοτρόπων ουσιών που αναζητούν οι χρήστες και τον ναρκωτικών. Αναφέρεται επίση στη σημασία που έχει η συλλογή στοιχείων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ζήτημα των τρίτων χωρών επίση. Γιατί το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι παγκόσμιο και διασυνοριακό. Επομένω, κατά την άποψή μου, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να δώσουμε τεχνική βοήθεια σε γειτονικέ χώρε και σε υποψήφιε προ ένταξη χώρε και για τη συλλογή πληροφοριών, αλλά και επίσης για την ανάπτυξη εργαλείων πρόληψης, αντίστοιχα με εκείνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο ε, να συνεργαστούμε με εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική γειτονία και την πολιτική της διεύρυνσης, να ε, τους δώσουμε τη δυνατότητα να ακούσουν τις παρουσιάσεις σας, τις λύσεις που έχει το κέντρο γιατί είναι ένα τομέα στον οποίο μπορεί να υπάρξει συνεργασία. γνωρίζω λίγο την κατάσταση με την Ουκρανία και με τη Μολδαβία και πιστεύω ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά. Τέλο. Αναφερθήκατε και σε κάποιε θετικέ εξελίξει, όπω για παράδειγμα τη μείωση των θανάτων από υπερβολική χρήση. Ε, εν μέρη ε, ε, εξαιτία και τη αύξηση τη πρόσβαση στα φάρμακα την, μετά την υπερβολική χρήση των οποίων Ωστόσο, το τελευταίο μου ερώτημα σχετίζεται ακριβώς με αυτό το, σύστημα, το νέο σύστημα της έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο είχαμε κρίνει και σιγά σιγά θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Θα ήθελα να μου δώσετε λίγες πληροφορίες για αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιουρέκ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα αυτά τα οποία είπατε, χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι μπορείτε να ανοιχνεύετε όλο και περισσότερες από αυτές τις νέες ουσίες. Ε, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ο ρόλος ε, της δικαιοσύνης. Ε, τι μπορείτε να μας πείτε για τον αριθμό αποφάσεων δικαστηρίων που αφορούν τα εγκλήματα περί ναρκωτικών, παραγωγή, διακίνηση, μικροδιακίνηση, χοντρική διακίνηση και πόσο σκληροί είναι οι δικαστές βλέπουμε κάποιον τρόπο αντιμετώπισης ε, των ε, ζητημάτων αυτών. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Και κάτι ακόμα από μένα θα ήθελα να πω. Στον ε, πρόεδρο ότι τοποθετήθηκε στο προηγούμενο θέμα. Το θέμα δεν αφορά τόσο την αναγκόμες, αλλά και το ότι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Μπορούμε να έχουμε πει μια ίση μεταχείριση πρέπει να παραιτηθούμε από αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γιούρεκ, όπως λέω, πάντα έχετε τέλειο timing γιατί θα πάρει τον λόγο πάλι η κυρία Γκόμες. Αλλά έχετε δίκαιο σε αυτό το οποίο λέτε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν απεκάλεσα κανέναν φασίστα. Είπα ότι η κατάσταση στην Ουγγαρία που βλέπουμε, όχι τώρα, εδώ και καιρό, έχει χαρακτηριστικά φασισμού. Ε, και δεν το ανακαλώ. Και βλέπω κάποιες ε, ε, κάποια συμπεριφορά των ε, αρχών που την θεωρώ φασιστική. Και επίσης ε, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαλβίνη που μιλούσε για τους Ρωμά και τους μετανάστες το περιγράφω ως φασιστικό και επιμένω σε αυτά. Είναι προσβλητικές οι λέξεις. Προσβλητική είναι αυτή η συμπεριφορά. Και θα έπρεπε να διακρίνουν αυτά, να τα διακρίνουν αυτά οι χώρε που τα γνώριζαν στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις ε, για εσάς. Και Για τα 37 cents τα οποία είπατε για τη χρηματοδότηση θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι πιο πιεστικές ανάγκες σας αυτή τη στιγμή. Είναι η χρηματοδότηση, είναι το προσωπικό. Γιατί βεβαίω και το προσωπικό πρέπει να πληρώνεται ή και τα δύο. Μετά για το θέμα μας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο για την Κίνα. Και αν υπάρχει κάποια ρύθμιση. Όταν η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είχε επισκεφθεί την Κίνα πριν από λίγα χρόνια για το θέμα αυτό, αντιμετωπίσαμε μια στάση απορριπτική από τις κινέζικες αρχές. Εντάξει, καταλάβαιναν ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν ήταν δικό τους πρόβλημα. Αυτοί το έκαναν εξαγωγή το πρόβλημα ήταν δικό μας. Έχει αλλάξει αυτή η στάση. Και κατόπιν βεβαίως είπατε ότι υπήρχαν κάποιες αλλαγές στους δρόμους ε, των εξαγωγών και στις διαδρομές των εξαγωγών. Και Βεβαίω οποιαδήποτε σχέση με την Βόρεια Αφρική και την σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και κατόπιν ε, υπάρχει και το θέμα της Λισαβόνα στην χώρα μου. Υπάρχει, έλεγχο, υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο των μικρών αεροδρομίων, ειδικά εκεί όπου υπάρχει μόνο ένας διάδρομος ε, προσγείωσης, που βεβαίως ε, είναι κάτι το πολύ ελκυστικό για τους παραδοσιακούς νοτιοαμερικανούς λαθροδιακίνητες. Δεν ξέρω αν έχετε εξετάσει τα θέματα της ε, Πορτογαλίας και αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, πληροφορίες. Τέλος, βλέπετε κάποια σχέση μεταξύ των ε, φοιτιών για καθαρά ιατρικούς σκοπούς και της αύξησης της παραγωγής ναρκωτικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχα ο άνθρωπο από τη Λισαβόνα. Και ο κ. Κόλιο, τέλο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες ανισχύτικες λεπτομέρειες ε, στην έκθεση αυτή. Αύξηση της παραγωγή στην Ευρώπη. Αύξηση ε, της παροχής ε, κοκαίνης. Όπως είπε και ο Διευθυντής, δεν είμαστε στην κορύφωση που είχαμε δει το 2014 όσον αφορά τις ε, νέες ουσίες, αλλά ούτως ή άλλως ε, έχουμε βρει νέες ψυχοτρόπες ουσίες όταν ψάχνουμε και θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε πέρσι και αφορούσε τους ανάψω από υπερβολική δόση Είχαμε μια τεράστια αύξηση πέρσι και παρά το γεγονός αυτό ε, που είχε τονιστεί στις σχέσεις με τις ίπα, εξακολουθούμε να έχουμε ε, υψηλό αριθμό υπερβολικών δόσεων και θα ήθελα να τονίσω το ότι υπάρχουν προβλήματα όταν ο κόσμος βγαίνει από την φυλακή και πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα όσο είναι στη φυλακή παρά το ότι γνωρίζουμε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Διευθυντή για την ποιότητα της έκθεσης και για την δουλειά που κάνουν στην υπηρεσία. Θα συμφωνήσω και εγώ κύριε Κοελιώνα με όλες τις ε, εκθέσεις αυτές. Το πρόβλημα είναι ότι για κάποιον λόγο και είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε ε, γιατί δεν έχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία το θέμα αυτό. Δηλαδή οι πολιτικοί παίζουν αυτά τα ζητήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι κακό παράδειγμα. Απλά ένα παράδειγμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μου μια σοβαρή συζήτηση για την κάναβη και την ιατρική της χρήση για παιδιά με επιληψή κτλ. το πρόβλημα είναι ότι σε αντίση με άλλους τομείς συχνά η συζήτηση δεν βασίζεται σε στοιχεία και βασίζεται σε πολιτισμικές και κοινωνικές συζητήσεις που έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό, ενώ σε άλλους ε, τομείς θα ήταν πολύ πιο σοβαρή η συζήτηση. Ελπίζω η Επιτροπή μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, τέσσερις βουλευτές που σε όλη την ε, συνεδρίαση για τον σεβασμό που έδειξαν στην έκθεση αυτή. Βλέπετε κύριε Κιουρεκ, ναι, εξαίρεσα τον ε, εαυτό μου. Θα το λέω γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό, γιατί να πω Τα στοιχεία στην έκθεση αυτή και στην προηγούμενη έκθεση είναι τόσο ανησυχητικά. Αλλάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία δραματικά. Και αν μου επιτρέπετε να σας δώσω άλλο ένα ανησυχητικό παράδειγμα, οποιοδήποτε αντιλαμβάνεται καθόλου τι είπα, και το τι συμβαίνει θα πρέπει να ξέρει το πώς τα ναρκωτικά μπορούν να αλλάξουν ολόκληρες ε, περιοχές. Και ακριβώς αυτό το θέμα για την αύξηση της χρήσης ε, των ναρκωτικών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά βεβαίω τα λέει ο κύριο Διευθυντή σε διάφορε εκθέσει και πρέπει να αποτελέσουν και συμπεράσματα για να περάσουμε στην πρόληψη. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τις ερωτήσεις τους και για τα καλά τους λόγια. Θα τα μεταφέρω και στους συναδέλφου μου. Ορισμένοι από αυτού μα παρακολουθούν και στη Λισαβόνα γιατί το, η έκθεση που σας παρουσιάζω είναι το αποτέλεσμα εργασίας πολλών ανθρώπων και στην υπηρεσία αλλά και επίσης με πολλούς άλλους, από πολλούς άλλους συνεργάτες που συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες και προσπαθούν να συνεισφέρουν στην ε, απάντηση που δίνουμε στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Το τονίσατε και εσείς πολύ καλά αυτό κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έρχομαι στις ερωτήσεις πρώτα απ' όλα του κυρίου Μπόνι Θα έλεγα ότι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συλλογή των πληροφοριών που σχετίζεται και με κάτι που είπε η κυρία Γκόμες αυτό ε, αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και αυτά είναι αρκετά στοιχεία, όμως θα χρειαστούμε επιπλέον πόρους, γιατί ε, και εσείς αναφέρθηκατε στην ανάλυση των δεδομένων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της επιδημιολογίας. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της μεταφοράς που ανέφερε ο κ. Μπόρνη. Ε, έχουμε μελέτες ε, τα τελευταία δύο χρόνια ε, online και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να καλύπτουμε όλο και περισσότερα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να προσταμοστούμε λοιπόν και θα έλεγα ότι ο λόγος είναι ο εξής. Πριν από 25 χρόνια ε, όταν δημιουργήθηκε το κέντρο, μας ζητήθηκε να παράγουμε εκθέσεις γιατί δεν υπήρχαν στατιστικά δεδομένα. Σήμερα έχουμε ε, στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται ε, τακτικά και με συνήθι τρόπο. Αυτά είναι η ραχοκοκαλιά των εικόνα που προσπαθούμε εμείς να συνθέσουμε, αλλά πρέπει να δούμε και την συνολικότερη ανάλυση τους. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια ενός έργου επιδημιολογίας και επίσης το δίκτυο Eurodem. Προσπαθούμε να και έχουμε πλέον συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα δίκτυα. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά εάν τελειώσει δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Γιατί εξάλλου δεν βρίσκονται αυτά τα δίκτυα στην εντολή του κέντρου. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι και το μόνο αίτημα και μόνο... Ε, το μόνο που θα ζητήσω για τον προπολογισμό την επόμενη χρονιά Έχουμε την μελέτη στα σχολεία. Θα θυμάστε ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα μοναδικό και χρηματοδοτήθηκε από την Σουηδία. Αποφασίστηκε από την Επιτροπή και τα κρατημέλη να ανατεθεί στο ECMDDA. Το αποδεχθήκαμε και με την υποστήριξη ε, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων που μας ε, έδωσε 310 εκατομμύρια ευρώ. Καταφέραμε να διεξάγουμε αυτή την έρευνα. Μία χρονιά όμως. Την επόμενη χρονιά δεν εγκρίθηκε το αντίστοιχο κοντιλέο από την DG Home. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα, ιδίω δεδομένου ότι θα αυξανόταν ο αριθμό των χωρών σε 30. Και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία. Αν λοιπόν θα μπορούσαμε για το 2019 να επανέλθει αυτή η χρηματοδότηση θα βοηθούσε πολύ. Έχει συζητηθεί το, ζήτημα της διεύρυνσης της εντολής της υπηρεσίας μας. Πιστεύω ότι ένα λύση θα ήταν να προβλεφθεί ξεχωριστό προπολογισμό για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία δεν αναφέρονται ε, στη, στη διακίνηση, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί πριν από 25 χρόνια. Τώρα, μιλώντα για τη διεθνή συνεργασία. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις υποψήφιες και πιθανώ υποψήφιες χώρες και έχουμε και αντίστοιχα κονδύλια για αυτή τη συνεργασία από τον υπο... προϋπολογισμό της Επιτροπής και το Ιανουάριο του 2019 θα ξεκινήσουμε και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με... με τι ε, γειτονικέ χώρε. Έρχομαι έτσι και στο ερώτημα τη κυρία Γκόμες μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα αυτό είναι ότι προβλέπεται πλέον ότι στο πρόγραμμα της Επιτροπής ότι θα μπορούμε να καλύπτουμε και τους χώρες που είναι όμορες προς τις γειτονικές μας χώρες. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι έχουν δημιουργηθεί νέες ε, διαδρομές για το, την κάναβη μέσω του Μαρόκου, μέσω της Λιβύης, της Αιγύπτου και άλλων τρίτων χώρων. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει σύνδεση ε, μεταξύ της διακίνησης ναρκωτικών, του τράφικινγκ και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όμως αυτή, αυτή η γνώση έχει έρθει χωρίς κάποια συστηματική μελέτη, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι υπόγειες διαδρομές και πώς μπορεί να προστατευθεί η Ευρώπη και να προστατεύσει τους πολίτες της. Αυτό είναι ένα κενό στη γνώση μας που θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε με το πρόγραμμα που σας ανέφερα. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι για όλες τις προτάσεις που μου κάνατε μάλλον θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να σας αποστείλουν ακόμα ένα email υπενθύμησης ώστε να απαντήσετε στην έρευνα που κάνουμε η οποία είναι ανοιχτή για τις επόμενες 6 ε, εβδομάδες. Θα θα σας δώσω τώρα κάποιες ορισμένες απαντήσεις και τις επόμενες, κύριε Μπόνη, ε, δύο εβδομάδες θα φροντίσω με τους συναδέλφους μου να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Γιατί πρέπει και να συντομεύσω. Έχουμε ε, μια σειρά δικτών για δικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Όμως αυτό αυτά μας δίνουν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Δεν γνωρίζουμε για παράδειγμα τι συμβαίνει με τις ποινές που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε κάποιες, ε, κάποια στοιχεία επίσης από τη Γενική Διεύθυνση Home για τις ελάχιστες ποινές. Θα σας τα αποστείλω και αυτά. Μιας και αναφερθήκατε όμως στις κατασχέσεις. Μπορώ να πω ότι αυτό παραμένει δύσκολο και πρόκληση στην Ευρώπη γιατί συνεχίζουμε να μην έχουμε στατιστικά στοιχεία για τις κατασχέσεις από, πολλές, από αρκετές χώρες και ιδιαίτερα μεγάλες χώρες. Δεν έχουμε στοιχεία ούτε για την ποσότητα, ούτε για την καθαρότητα, ούτε για το είδος των ουσιών. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε αυτό με διμερείς ε, επαφές, ε, επικοινωνώντας ε, με τα κράτη-μέλη και θα συζητήσουμε επίσης το ζήτημα αυτό με την, το Διοικητικό Συμβούλιο στη Λισαβόνα την επόμενη εβδομάδα πάλι. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε περισσότερα εδώ Το πρόβλημα δεν είναι τόσο να δημιουργήσουμε νέους δείκτες και να ζητήσουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά πώς θα αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Για να έρθω τώρα στη ερώτημα της κυρίας Γκόμες, που εν μέρη νομίζω ήδη το απάντησα, μία από τις πρώτες δηλώσεις που έκανα μετά την, τον εκλογή μου, είχα πει ότι θα προσπαθήσω να είμαι προγραμματιστής και λογικός και δεν ζήτησα αύξηση του προπολογισμού γιατί έπρεπε πρώτα απ' όλα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της υπηρεσίας μας και να προσφέρουμε περισσότερη υπηρεσία στις αξία με τα χρήματα που έχουμε. Και θα έλεγα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όμως, θα έλεγα, το 2019 αν θα μπορούσαμε να ε, επανακτήσουμε αυτές τις 310.000 που χάθηκαν, νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει να κλείσουμε το χάσμα που θα υπάρξει ανάμεσα στο σήμερα ή το, του χρόνου και το χρονικό σημείο που θα έχουμε το νέο κανονισμό. Ε, κατά τα άλλα, ε, μπορώ να σας ενημερώσω γραπτός για τις υπόλοιπες ερωτήσεις για τα αεροδρόμια. Με ρωτήσατε επίσης για την Κίνα. Μου το είπε το πρωί ο κύριος Διπχέ μάλιστα ότι όταν το επιθυμεί η Κίνα μπορεί να ελέγχει πολύ αποτελεσματικά. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις ουσίες. Πάντως, ορισμένες από τις ψυχοτρόπους ουσίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, όμως αυτό δεν αρκεί και επίσης διαπιστώνουμε ότι η μεταφορά, διακίνηση αυτών των ουσιών γίνεται μαζικά και φανταστείτε τον αριθμό των κοντέινερ τα οποία πρέπει να εκτελονιστούν και περνούν από τις διαδικασίες σε ένα λιμάνι όπως το Ρότερνταμ. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς τους απαιτούμενους ελέγχους. Αναφερθήκατε στη σύνδεση με την εμπορία ανθρώπων. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνάντηση σχετική και ε, συμφωνήθηκε στο επίπεδο όλων των γενικών διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Home και των σχετικών υπηρεσιών να ασχοληθούμε και να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ μας στην αντιμετώπιση του τράφικινγκ. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τον κύριο Κοέλιο για τις, τα, τα καλά σας λόγια Γνωρίζω ότι ίσως να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, την ερώτηση της κυρίας Γκόμες για παράδειγμα, και θα κλείσω με αυτό γιατί συνδέεται με αυτό που είπε ο Πρόεδρος, που, είναι, που έχει σχέση με την φαρμακευτική χρήση της κάναβης και τις διάφορες πολιτικές που βλέπουν να υιοθετούνται στα Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις και ε, να ε, συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία, ουσιαστικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην ε, διαδίδουμε στερεότυπα. Θα έλεγα ότι συνεισφέραμε στην προσπάθεια να καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι προκλήσεις όταν γίνεται μια προσπάθεια νομιμοποίησης ορισμένων χρήσεων της κάναβης και σε κάποιες χώρες. Είχαμε μια σχετική έκθεση δημοσιοποίηση πριν από λίγες εβδομάδες. Θα δω επίσης με τους συναδέλφους αν μπορούμε να σας στείλουμε και μία έκθεση την οποία προετοιμάζουμε που είναι μία μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας για την ε, ιατρική χρήση της κάναβης και των παραγόγων ουσιών από την κάναβη. Θα δω αν μπορούμε να σας το στείλουμε έτσι ώστε να έχετε περισσότερες αντικειμενικές πληροφορίες στα χέρια σας. Προετοιμάζουμε επίσης και ακόμα μια έκδοση μέχρι το τέλος της χρονιάς που θα περιγράφει την κατάσταση με αγορές ε, κάναβης οι οποίες έχουν ρυθμιστικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Θα έχουμε και αποστολή στη Λισαβόνα, στο MCDDA, τον Οκτώβριο. Και να σας πω με την ευκαιρία ότι η έδρα του οργανισμού σας βρίσκεται σε μια εξαιρετική πόλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και όλους τους συναδέλφους σας που βλέπουν τη συνεδρίαση μας μέσω του ίντερνετ, στο webstream. Το τα, συνεχάρει ο κύριος Κοέλιο με τρόπο πολύ ομορφότερο από ό,τι θα μπορούσα εγώ ποτέ να το κάνω. Ίσως να το έχω πει και παλιά, θα ήθελα πριν τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου με τους συναδέλφους που έχουν ιδιαίτερε γνώσει και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ζήτημα των ψυχοτρόπων ουσιών και των ναρκωτικών, να οργανώσουμε κάτι, ε, ίσως κάποια εκδήλωση περισσότερο εστιασμένη σε αυτό το θέμα. για να ακούσουμε ε, ε, τα, τα ζητήματα αυτά που, και τα στοιχεία που αναδεικνύεται. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που τα γνωρίζουν τα θέματα αυτά, όπω ο κ. Μπον και άλλοι. Θα ήθελα και πάλι να σα ευχαριστήσω και θα κλείσουμε τη σημερινή μα συνεδρίαση εδώ. Επόμενη συνεδρίαση αύριο το πρωί. Καλό απόγευμα. Thank you very much. Thanks. Uh, I will check if we can have first draft.